Good morning. I will speak in Spanish. Καλημέρα, θα μιλήσω ισπανικά. Bueno, vamos a abrir la sesión. Άρχεται η συνεδρίαση. Βάσει του άρθρου 14, παράγραφος 1 του κανονισμού, θα προεδρεύσω ως αντιπρόεδρος, δεδομένου ότι ο απερχόμενος πρόεδρος απουσιάζει. Να σας πω ότι σκοπός της συνεδρίασης είναι η συγκρότηση ε, του Προεδρίου, εκλογή του Προέδρου και των τεσσάρων αντιπροέδρων, βάσει του άρθρου 204 του ιστορικού κανονισμού. Ενημερίθηκα για τους αναπληρωτές που συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Αν υπάρξει κάποια αλλαγή, οι πολιτικές ομάδες μπορούν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο πριν από την ψηφοφορία. Θα ήθελα να ζητήσω από τη Γραμματεία να ε, επιβεβαιώσει ότι υπάρχει απαρτία προκειμένου να είναι έγκυρη ψηφοφορία και να σας πω ότι βάσει του άρθρου 208 η απαρτία είναι το 1 τέταρτο των μελών της Επιτροπής, δηλαδή 19 μέλη. Υπάρχει απαρτία. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω τους υποψηφίους για την Προεδρία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ο υποψήφιος πρέπει να οριστεί από μια πολιτική ομάδα ή από το 25% των μελών της Επιτροπής, 4 μέλη, συγγνώμη, το 5%, 4 μέλη. Ε, ο κύριος Πρέδα έχει το λόγο, έχει οριστεί ο κύριος Μακάλιστερος υποψήφιος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν πω δύο για την πρόταση που έγινε από την πολιτική μας ομάδα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο ε, της Επιτροπής, ε, τον κύριο Έλμαρ Μπρόκ, για τις δραστηριότητές τους. Δυστυχώς σήμερα πουσιάζει, αλλά ε, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω όχι μόνο για τα όσα έκανε ως πρόεδρος της Επιτροπής μας αυτά τα δυόμιση χρόνια, αλλά επίσης και για τις δραστηριότητές του. Να υπενθυμίσω ότι εξελέγει το 1980 εδώ στο Κοινοβούλιο. Οι δραστηριότητές του, η εργασία του είναι απόλυτα αναγνωρισμένα και θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Maintenant, euh, la proposition... Τώρα η πρόταση της πολιτικής μας ομάδος για πρόεδρο της Επιτροπής μας είναι ο κύριος Ντέιβιτ Μακάλιστερ. Πρόκειται για έναν συνάδελφο ο οποίος ε, από το 1998 ε, είναι ευρωβουλευτής, ήταν συγγνώμη βουλευτής ε, ε, στην ε, χώρα του. Το 2014 ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το γνωρίζετε γιατί ήταν ε, εισηγητής για τη Σερβία, όπου επέδειξε και το ευρωπαϊκό του αίσθημα, την πολιτική του ευφυΐα και τον υποστηρίζουμε για πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη επόμενα δυόμιση χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από τον υποψήφιο, από τον κύριο Ντέβιτ Μακάλιστερ, να αποδέχεται την υποψηφιότητα. Ναι. Ο υποψήφιος λοιπόν πληρεί τις προϋποθέσεις, είναι μέλος της Επιτροπής, έχει υπογράψει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες, προτείνω να εκλεγεί διαβοής ο υποψήφιος, ο οποίος μπορεί να έρθει εδώ να αναλάβει τα εννέα. Liebe Kolleginnen und Kollegen, συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Για μένα είναι μια ιδιαίτερη τιμή να προεδρεύω αυτής της Επιτροπής για τα επόμενα δυόμιση χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ε, ψήφο σας και θα ήθελα επίσης να πω ορισμένα προσωπικά λόγια ευχαριστίας ε, προς τον Έλμαρ Μπρόκ, ο οποίος ε, σήμερα δεν είναι στις Βρυξέλλες γιατί ήθελε να τιμήσει τον Ρόμαρ Χέρτσοκ, τον πρόεδρο της Γερμανίας, ο οποίος ε, πέθανε και γίνεται σήμερα η τελετή στο Βερολίνο. Είναι ο παλαιότερος ε, βουλευτής εδώ ε, και 37 χρόνια και παραμένει βουλευτής του Ευρωκοινοβουλίου και θα συμβάλλει με την εξαιρετικά πολύτιμη εμπειρία του. Θα ήθελα να διασφαλίσω να βεβαιώσω τα μέλη της Επιτροπής ότι θα ήθελα να στηριχτώ σε μια πλατιά συνεργασία και θα ήθελα να απευθυνθώ προς τους συντονιστές αλλά όχι μόνον και προς τα μέλη ε, και τα αναπληρωματικά μέλη αυτής της Επιτροπής εάν έχετε κάποια ερωτήματα ή έχετε κάποιες προτάσεις μη διστάσετε να απευθυνθείτε άμεσα σε μένα ή τους αντιπροέδρους και τη γραμματεία θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε μια συμφωνία τους ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστοσύνη σας και την, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και δική μου πολιτική ομάδα που με πρότεινε. Τώρα, με την ε, γραμματεία συζήτησα ε, και είπαμε ότι για πρακτικούς λόγους θα γίνει η συνεδρίαση στα αγγλικά κατ' ουσία γιατί αυτό διευκολύνει την επικοινωνία για όλους μας. Γι' αυτό θα περάσω τώρα στα αγγλικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να, σας, ε, να περάσουμε στο επόμενο σημείο της σας διάταξη, δηλαδή την εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου. Ε, και πάλι υποθέτω ότι θα, θα πρέπει να ζητήσω τις ε, πολιτικές ομάδες να αποβάλουν τις προτάσεις τους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω την υποψηφιότητα του Άντες Χριστιστον, ενός ευρωβουλευτή από τη Δανία, ο οποίος ε, πραγματικά είναι απολύτως ικανός για αυτή την ε, θέση. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω τον Άντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες προτάσεις. Όχι. εφόσον είστε ένα νέος ε, συνάδελφος σε αυτή την Επιτροπή, ίσω θα θέλατε να πείτε μερικά λόγια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που με προτείνατε για αυτή τη θέση. Είμαι νέο συνάδελφος σε αυτή την Επιτροπή, αλλά πραγματικά ανέμενα με ανυπομονησία να συνεργαστώ μαζί σας ε, και θα προσπαθήσω, εάν δεν παρίσταται ο Πρόεδρος, να ε, συντονίσω τις εργασίες με έναν αμερόληπτο τρόπο και είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με όλους σας για να ε, εκπληρώσουμε το πολιτικό έργο το οποίο καλούμεθα να πράξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Διαβοής μπορούμε να επικαιρώσουμε την εκλογή. Περ, παρακαλώ διαβοής. Ωραία λοιπόν. Μπορείτε κι εσείς ε, να έρθετε εδώ στο Προεδρείο και στη συνέχεια θα περάσουμε στο επόμενο σημείο την εκλογή του Δευτέρου Αντιπροέδρου αυτής της Επιτροπής και πάλι θα ήθελα να ζητήσω να υποβάλλετε τις προτάσεις σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η πολιτική μου ομάδα, η ΚΟΕ, θα ήθελε να προτείνει τον ε, Χαβιέ Κούσο, τον ε, πραγματικά ε, αξιόλογο συνάδελφο που απολαμβάνει τις εμπιστοσύνη ολόκληρης της πολιτικής ομάδας και τα προηγούμενα δυόμιση έτη επετέλεσε το αξίωμά του πραγματικά με μεγάλη αξιοπιστία και ικανότητα. Μπορούμε να τον εμπιστευτούμε και θα ήθελα να επικαιρώσετε την εκλογή του ως Δευτέρου Αντιπροέδρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Λέζινγκ. Ε, και μπορούμε τώρα να περάσουμε και πάλι στο διορισμό διαβοής. Παρακαλώ. Ε, κατά, αποχές, ωραία λοιπόν, επικαιρώνεται η εκλογή, θερμά συγχαρητήρια. Και τώρα θα περάσουμε στην εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου. Παρακαλώ κυρία Φλέκενστάιν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αντικριστέ. Ο, ο, ο συνάδελφος εκτεξιών μου είναι γνωστός στην Επιτροπή και είναι ιδιαίτερα ε, δεσμευμένος, επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο ως πρόεδρος της Επιτροπής Συνεργασίας με την Μολδαβία και είναι δραστήριο σε πολλούς τομείς και είναι απολύτως αξιόπιστος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φλέκενστάιν. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Όχι, άρα μπορούμε και εδώ η διαβοής να ε, διορίσουμε τον, τρίτο αντιπρόεδρό μας. Ε, και σε εσά εύχομαι θερμά συγχαρητήρια και θα περάσουμε τώρα στον τέταρτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής, και εδώ παρακαλώ να υποβάλλετε τις προτάσεις σας. Κρίστιαν Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική μας ομάδα προτείνει για τη θέση αυτή το συνάδελφο Ντόμπραφ Κρισχαφκουίτσα, ο οποίος ε, ε, υπήρξε ήδη αντιπρόεδρος της Επιτροπής, έχει μια πολιτική εμπειρία, είναι πολύ παλαιό μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών ε, Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες ε, προτάσεις. Όχι. Ντουμπράφκα Ζούιτσα, υπέρ. Διαβοής. Ωραία λοιπόν, συγχαρητήρια και καλή συνεργασία. Παρακαλώ, αγαπητέ συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από δέκα χρόνια ε, θητείας εδώ ως Αντιπροέδρου στην ΑΦΕΤ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ και θα πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι ότι είναι μεγάλη μου τιμή και ελπίζω ε, να έχουμε και μια ευχάριστη ε, θητεία μαζί. Right, we're at the end of... Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το πρώτο τμήμα της συνεδρίασής μας και θα συνεχίσουμε στις 9.30, δηλαδή σε 7 λεπτά για μια κοινή συνεδρίαση με τους συναδέλφους από την ΤΕΒΕ.

Θα, θα, δούμε, θα δούμε πώς θα πάει τώρα η δουλειά. Εντάξει, το αργότερο δούμε... 10.30 να... Ναι, ναι, θα όχι, θα δούμε πιο νωρίς. Για να προλάβουμε να πάμε και. Δεν ξέρω, θα, θα, θα δω, πώς θα, πάει. Πώς θα κυλήσει και εδώ η διαδικασία. Δεν σε κανένα μισό, αλλά θα φύγουμε, γιατί δεν έχει... Μπορείτε να κάνετε παρέμβαση εδώ. Θέλω να προλάβουμε να... Δεν, ξέρω, δεν προλάβουμε. Ladies and gentlemen, dear colleagues, Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε τώρα την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης. Βέβαια, να καλωσορίσω και τη συνάδελφο κυρία Μακάβων, πρόεδρο της Επιτροπής. Αρχικά να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι να περάσουμε στο σημείο 2, ας κάνω την εξή ανακοίνωση. Αγαπητοί συνάδελφοι τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, να γνωρίζετε ότι αύριο θα έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση τη ε, αντιπροσωπεία ε, προ την ε, Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Ολομέλεια με τον κύριο Λούί Αλμάντρο. Όλα τα μέλη τη Επιτροπής ΑΦΕΤ προσκαλούνται να παρευρεθούν και η συνεδρία θα λάβει χώρα αύριο από τις 5 έως τις 6 το απόγευμα στο κτίριο Αλτιέρος Πινέλη στην αίθουσα 1Ε2. Αυτή ήταν η ανακοίνωσή μου. Λοιπόν, περνούμε τώρα στο σημείο 2 σε σχέση με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και τον ρόλο της υπηρεσίας ευθετικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα εξετάσουμε λοιπόν αυτή την ε, ιδιαίτερα επίκαιρη ε, έκθεση ίδια πρωτοβουλία με 547 τροπολογίες παρακαλώ για αυτή την έκθεση, για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα και 37 συμβαστικέ τροπολογίε. Έχουν τύχει διαπραγμάτευση και έχουν συμφωνηθεί. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε στι 31 Ιανουαρίου το απόγευμα στι Βρυξέλλε. Αν συμφωνείτε και εσεί, κυρία Μακάβων, μπορούμε να δώσουμε τώρα το λόγο στου ε, συνεισηγητέ η κυρία Ελένα Βαλενσιάνο και ο κύριο Δία Δεμέρα. Ποιο θα ήθελε να πάρει το λόγο πρώτος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώ ήλθατε και σε συγχαρητήρια για την εκλογή σα. Αυτή είναι η τελευταία συζήτηση που κάνουμε για αυτή την έκθεση η οποία, όπως εξήγησε ο Πρόεδρος, είναι μια κοινή έκθεση μεταξύ ε, Επιτροπών ΑΦΕΤ και ΝΤΕΒΕ. Θα ήθελα καταρχάς ε, να ευχαριστήσω ιδιαίτερος ε, τον συνεισηγητή μου, τον κύριο Διαθτεμέρα, ο οποίος είναι εισηγητής εκ μέρους Επιτροπής Ανάπτυξης για την εξαιρετική συνεργασία κατά την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Πρόκειται για μια κοινή έκθεση και όπως γνωρίζετε ε, βάσει του άρθρου 54 όπως προβλέπετε, ορισμένες φορές μπορεί να γίνει και κόλαση. Αυτή τη φορά ήταν ακριβώς το αντίθετο και χάρηκα που μπορέσαμε να ε, φτιάξουμε αυτή την έκθεση από κοινού μεταξύ των ε, δύο συγητών. Να ευχαριστήσω επίσης και τους σκιώδεις συγητές οι οποίοι βοήθησαν ιδιαίτερα και έτσι είχαμε πολύ ευρεία συνένεση για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το οποίο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποστείλει ένα πάρα πολύ ισχυρό και σαφές μήνυμα. Ε, γι' αυτό λοιπόν είναι και πάρα πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε όλοι. Το πρώτο σχέδιο κειμένου είχε περίπου 550 τροπολογίες και οι δύο εισηγητές ε, ασχοληθήκαμε με την εικόνα συμβιβαστικών τροπολογιών ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες φωνές. Για μας η επίτευξη της συνένεσης ήταν ένα από τα ε, στοιχεία τα οποία αποτέλεσαν προτεραιότητα κατά την εκπόνηση της έκθεσης. Έχουμε 37 ε, συμβαστικές τροπολογίες ε, και έτσι θα ενσωματωθούν πάνω από 230 τροπολογίες και διαθέτεται και την τελευταία εκδοχή αυτών των ε, τελευταίων συμβαστικών τροπολογιών. Ελάχιστες αλλαγές είχαμε. Έγινε μια συνεδρίαση σχεδόν εισηγητών σε τεχνικό επίπεδο. Η έκθεση αυτή, κύριε Πρόεδρε, αντιμετωπίζει μια εξωτερική πτυχή η οποία μέχρι τούδε αποτελούσε πολύ μεγάλο έλλειμμα στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο τομέας της μετανάστευσης ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα των Υπουργών Εσωτερικών και ε, έτσι ε, καταφέρνουμε να έχουμε ένα πιο ανοιχτό πρίσμα το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε μια πιο ε, πλήρη πολιτική σε εξωτερικά θέματα. Μέσω του νέου πλαισίου εταιρική σχέση, τα λεγόμενα compact, καταφέρνουμε σιγά σιγά να αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε και βέβαιοι ότι θα ακολουθήσουμε τη σωστή άγουσα. Συνειδητοποιούμε πόσε δυσκολίε έχει ε, όλο αυτό το θέμα. Γίνονται προσπάθειε και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από πλευρά Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, ενώπιον ενό Συμβουλίου, ενώπιον κάποιων εθνικών κυβερνήσεων που, για να το πω διπλωματικά, δεν έχουν αρκετή ευαισθησία για να αντιμετωπίσουν και ίσως και όχι αρκετή ευφυΐα για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως. Θα ήθελα τώρα να σταθώ πολύ γρήγορα σε κάποιες βασικές ιδέες οι οποίες αποτελούν ε, πυλώνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και περιλαμβάνονται και στις συμβαστικές τροπολογίες. Καταρχάς, τα δικαιώματα και αξιοπρέπεια των ατόμων, είτε πρόκειται για πρόσφυγο, για ε, ε, αισθητούντες άσυλο ή απλούς παράνομος μετανάστευση δεν θα πρέπει να μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Δεύτερον, οι μεταναστευτικές ροέ δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως απειλή. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που τα αντιλαμβανόμαστε και θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα είναι επωφελές και για τις δύο πλευρές, και για τους ανθρώπους που έρχονται στι χώρε μα αλλά και για μα. Πρόκειται για μία μάχη που δεν θα πρέπει να χάσουμε εμεί ω δημοκράτε και θα πρέπει να δώσουμε χωρί συμπλέγματα ενώπιον μια άκρα δεξιά η οποία είναι ξενοφοβική και ακραία σε όλο τον κόσμο. Τρίτον, η πολιτική συνεργασία μα θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να δώσει απαντήσει στι πολλαπλέ αιτίε των ε, μεταναστευτικών φαινομένων, ώστε η μετανάστευση να είναι μία επιλογή και όχι μία υποχρέωση. Τέταρτον, η βοήθειά μας θα πρέπει να είναι άνεφόρον και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να επιτύχουμε συνεργασία τρίτων χωρών σε θέματα επανεισδοχής ή ελέγχου των ε, μετακινήσεων. Πέμπτον, εάν πραγματικά πρέπει να σταματήσει η διακίνηση ανθρώπων και να σταματήσει ο πόνος αυτών των χιλιάδων ανθρώπων που δεν έχουν τίποτα άλλο να χάσουν παρά μόνο τη ζωή τους, θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλείς και νόμιμες οδοί μετανάστευσης, για παράδειγμα μέσω ανθρωπιστικών θεωρήσεων. Και να έχουν και μια άλλη επιλογή, το να μην ξεκινήσουν δηλαδή ένα ταξίδι αυτοκτονίας μέσω της Μεσογείου θάλασσας. Έκτον, θα πρέπει να σταματήσουμε να περιμένουμε μια πραγματική πολιτική μετανάστευση. Πρέπει να υλοποιηθεί και πρέπει να βασίζεται στην πολιτική τη αλληλεγγύη και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έβδομον, μια ένωση η οποία έρχεται σε αντίθεση με τι πολιτικέ τη, ε, στι ίδιε τι αξίε, είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να τηρήσουμε τι δεσμόψει μα, γιατί αλλιώ είμαστε καταδικασμένοι να αποτύχουμε ε, όχι μόνο στα θέματα της πολιτικής και της μετανάστευσης και στους πρόσφυγες, αλλά σε παγκόσμιο πλαίσιο. 8. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να μείνει στο περιθώριο κατά το σχεδιασμό των διαφόρων δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα τα λεγόμενα Migration Compacts και τις συνέπειες που υπάρχουν για τον προπολογισμό στα θέματα αυτά. Αυτά είναι τα κεντρικά στοιχεία του μηνύματος που θέλουμε να αποστείλουμε και όλες οι πολιτικές ομάδες συνεργάστηκαν ε, και συμφωνούμε από αυτού. Υπάρχουν ε, κάποια θέματα ε, τα οποία δεν μπόρεσαν να συμπεριληφθούν στις συμβαστικές προτάσεις και έχουν σχέση με συγκεκριμένες περιπτώσεις και δύσκολες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα την Τουρκία ή το Αφγανιστάν. Πρέπει να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανησυχεί σοβαρά για μια νέα τάση που φαίνεται να εμφανίζεται σε σχέση με το μοντέλο το οποίο ε, προκύπτει ε, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία με την Τουρκία. Μπορεί να υπάρξει και μια αντίστοιχη συμφωνία με τη Λιβύη και δεν ξέρω κατά πόσον θα το ε, αποδεχτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο εγγύς μέλλον ε, τα διάφορα ε, compact θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικά ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε προς αυτή τη σωστή κατεύθυνση και να εδραιώσουμε την πολιτική μας. Δεν θα ήθελα να καθυστερήσω άλλο τη συζήτηση. Είμαι στη διάθεση των συναδέλφων για οποιοδήποτε ζήτημα διευκρίνηση όσον αφορά τις συμβαστικές προτάσεις και σας ευχαριστώ όλους για την πολύ επικοδομητική σας στάση και την πολύ ευφυή στάση που επιδείξετε και θα συμπεριλάβω και ε, τη γραμματεία βεβαίως ε, στις ευχαριστίες μου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε αγαπητή συνάδελφα. Και τώρα ο λόγος του κύριο Δίας Δεμέρας, ενησυχητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε. Θα πω λίγα πράγματα. αλλά θα ήθελα να πω το εξής, ε, να τονίσω την ε, σημασία αυτής της συμφωνίας όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 55 και μου έδωσε την ευκαιρία να επικαιρώσω την, ε, να, την ποιότητα της εργασίας της κυρίας Βαλενθιάνα ως πολιτικού και ως προσωπικότητα συνενετικής πρόθυμης να ανοίξει το διάλογο. Ε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ, Έλενα. Είναι εξαιρετικά πολύτιμο το έργο σου. Ε, και θα ήταν δίκαιο να ευχαριστήσουμε και τους Σκιώδης για το έργο σου που μας βοήθησαν να καταλήξουμε ε, μεταξύ των σε, στους, στις συμβαστικές ε, τροπολογίες δεν ήταν εύκολο το έργο και συνέβαλαν πραγματικά με μεγάλο επαγγελματισμό καθώς και τα μέλη της Γραμματείας των Επιτροπών και οι συνεργάτες μας οι πιο άμεση. Ε, η δική μου πολιτική ομάδα στηρίζει όλες τις συμβαστικές τροπολογίες. Πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα, σημαντικό ούτως ώστε ε, μαζί με την ε, ομάδα που υποστηρίζει, που εκπροσωπεί η Ελένα, ε, προσδίδει μια μεγάλη αξία σε ένα θέμα τόσο πολύπλοκο όπως είναι το θέμα των μεταναστευτικών ροών και η διασύνδεση του θέματος αυτό με την εξωτερική, με την υπηρεσία εξωτερικής δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και του, του για να μην ε, επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν, θα ήθελα να δώσω έμφαση ε, σε, ορισμένα ερωτήματα. Την σημασία που έχει η διασύνδεση της ε, κινητικότητας με την αλληλεγγύη. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Επίσης είναι ουσιώδες να συνδέσουμε την ε, μετανάστευση και την ε, ανάπτυξη. Είναι εξίσου σημαντικό να λάβετε υπόψη σας ότι σκεμμένα δώσαμε την έμφαση σε θέματα όπως είναι η ανθρωπιστική βοήθεια, το ζήτημα του φύλου και οι ιδιαίτερα ευάλωτε ομάδε και όλα αυτά σύμφωνα με, το, με, την, ε, με, την, ε, με το πνεύμα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι αναγκαίο να, πούμε, να τονίσουμε το έργο των περιφερειακών και υποπεριφερειακών ε, οργανώσεων Ένα θέμα για μας αδιαμφισβήτητο είναι ο ρόλος, ο ανατικός ρόλος που παίζει η κλιματική αλλαγή, θέμα το οποίο βεβαίως έχουν θέσει και άλλοι οι οποίοι ε, ε, είναι, δεν είναι ανταΐσεις με το θέμα αυτό. Τώρα, όσον αφορά τις νόμιμες ε, οδούς και σε σχέση με την ανθρωπιστική δράση, σε σχέση με πολιτικά ζητήματα τα οποία δεν έχουν ε, επιληθεί και έχουν προσλάβει δραματικές ε, διαστάσεις, η μη συμφωνία με την Τουρκία και βεβαίως ο πόλεμος στη Συρία. Και δεν θα ήθελα να παραλείψω τα, το ζήτημα των χρηματοδοτικών και για να καταλήξω θα ήθελα να πω ότι η μετανάστευση αποτελεί δικαίωμα και αυτό το τονίζουμε στην έκθεσή μας. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την ε, συνεργασία τους, για την ολοκλήρωση αυτής της έκθεσης και όπως και η Ελένα, θα ήθελα να πω ότι βρίσκομαι στη διάθεσή σας για τυχόν ε, ερωτήματα. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο συναδέλφους. Τώρα μπορούμε να αρχίσουμε τη συζήτηση. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους ε, σκιώδεις εισηγητές, τουλάχιστον σε όσους ε, παρίστανται. Η κυρία Λόχμπιλερ είναι η πρώτη ομιλήτρια από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας και από τη δική μας ε, πολιτική ομάδα ε, και περιμένουμε μεγάλη προσμονή να συνεργαστούμε μαζί σας. Όσο εσκιώδης συγγήτρια θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, δύο συνεισηγητές για την εξαιρετική αυτή και διαδικασία και με που έχει και ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι σημαντική η έκθεση, είναι το πρώτο βήμα για το Κοινοβούλιο να αντιμετωπίσει και να εξετάσει τη σημασία της βελτίωσης ε, της συνοχής της συνεργασίας με τρίτες χώρες για τη μετανάστευση με σκοπό την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, τη δέωση επιμέλεια. Ε, όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ενσωματώνονται σε πιθανές συμφωνίες με χώρες διέλευσης ε, και προέλευσης με σκοπό την κοινωνική συνεργασία τελικά. Ιδίω η χρηστή διακυβέρνηση, αναπτυξιακή στόχη για τα ευρωπαϊκά, τους ευρωπαϊκούς πόρους θα πρέπει να ε, προωθηθεί ω ε, τμήμα των μεταναστευτικών συμφωνιών με τρίτες χώρες. Τα πρόσφατα παραδείγματα όπω είναι η συμφωνία με την Τουρκία και με το Αφγανιστάν ή η άτυπη ε, πρόσφατη συμφωνία με το Μαλί δείχνουν ότι η βελτίωση της συνεργασίας με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης δεν ε, έχει την επαρκή διαφάνεια και όλο ένα και περισσότερο εστιάζει στην αποτροπή της παράτυπης ε, μετανάστευσης και στην αύξηση του αριθμού των επιστροφών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και χωρίς να αντιμετωπίζει τις αιτίες, τη ρίζα δηλαδή του προβλήματος, ε, να αντιμετωπίσει δηλαδή τι αιτίε που οδηγούν κάποιον στο μεταναστεύσει. Αυτή η ανεπαρκή εστίαση στα ανθρώπινα δικαιώματα ε, οδηγεί ε, όλα για περισσότερε περισσότερο σε ανησυχητικέ παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην κακομεταχείριση των μεταναστών στα κέντρα υποδοχή και σε έλλειψη εποπτείας όταν υπάρχουν αυτές οι παραβάσεις είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε την αξία της σημασίας ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αυτής και να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Όσο εκ τούτου θα είναι απαραίτητο ε, να δώσουμε περισσότερες ε, εγγυήσεις και την δικλείδες ασφαλείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ε, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και με το μηχανισμό προστασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διασφαλίσουμε την κοινοβουλευτική εποπτεία και δημοκρατική εποπτεία στον τομέα της συνεργασίας ε, και ε, μεταναστευτικής διαχείρισης. Οι άτυπες συμφωνίες όπως το Joint Way Forward μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφγανιστάν και η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία δεν θα πρέπει να αποτελέσουν το πρότυπο συνεργασία σε τρίτε χώρε στον τομέα τη μετανάστευση και διαχείριση ροών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δραματίσει ισχυρό ρόλο ε, στη δημοκρατική εξέταση και εποπτεία αυτών των συμφωνιών και η κοινοβουλευτική εποπτεία δεν θα πρέπει να αποφεύγεται. Και υπενθυμίζουμε ότι η αναπτυξιακή συνεργασία θα πρέπει να έχει ως στόχο την εξάλληψη της φτώχειας και θα πρέπει με αυτή την έκθεση να τονίσουμε ότι ο μοναδικός βιώσιμος τρόπος είναι ένα πιο ανθρώπινο πλαίσιο συνεργασίας με τέτοιες χώρες, διατηρώντας την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια στις μεγάλες ε, μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές και να προωθούμε την ισομερή κατανομή των ε, βαρών και να έχουμε και ασφαλείς και νόμιμες οδούς μετανάστευσης. Ελπίζουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά ε, πιο αναλυτικά ε, στις κοινέ τροπολογίες, τις περισσότερες τις οποίες μπορούμε να στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε πολύ. Α, ευχαριστούμε κυρία Λόχπιλερ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Βερζιά από την ΚΟΕ. Oui, merci, monsieur Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, συγχαρητήρια καταρχήν για την εκλογή σας. Θα ήθελα να συγχωρήσω τον συνάδελφο Μικέλ Ορμπάν και γιατί θα μιλήσω τόσο ως εκπρόσωπος της ΚΟΕ ως και εισηγήτρια της Επιτροπής ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο ε, συνεισηγητές και τους Κιώδης και θεωρώ ότι η έκθεση αυτή εντάσσεται στη συνέχεια των εκθέσεων που εγκρίναμε τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια για τη μετανάστευση ε, σε τρίτες ε, χώρες και υπάρχουν ε, εδώ πολλά στοιχεία στις συμβαστικές τροπολογίες τα οποία αντανακλούν, εάν θέλετε, τις, εκείνες τις προηγούμενες εκθέσεις και θα ήθελα να επιμείνω σε ορισμένα σημεία τα οποία είναι σημαντικά για τη ΛΥΜΠΕ και στα οποία δεν δίνεται ακριβώς η ίδια έμφαση στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Όσον αφορά τους απάτριδες, το θέμα αυτό νομίζω ότι δεν αντιμετωπίζεται αρκετά στην έκθεση. Η ΛΥΜΠΕ όμως δίνει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό γιατί πρόκειται για ένα όλο και πιο σημαντικό θέμα και το οποίο συνδέεται με τις μεταναστευτικές ροές και ιδιαίτερα ε, με το, το ζήτημα των παιδιών, τα οποία είναι δύσκολο να αναγνωριστούν αυτή τη στιγμή έχουν καταλήψει τη χώρα τους. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επιμείνω είναι πέρα από αυτό το οποίο αναφέρεται στις συμβαστικές τροπολογίες, η αξιολόγηση και ο έλεγχος των κονδυλίων τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλες αυτές τις πολιτικές γιατί έχουμε την εντύπωση ότι τα ζητήματα αυτά υπεκφεύγουν του ε, ελέγχου του Ευρωκοινοβουλίου και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να επιμείνουμε στην ανάγκη να αξιολογούμε το σύνολο των κονδυλίων ε, στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής και σε σχέση με δεχόμενες ε, αποκλήσεις που μπορεί να υπάρξουν όσον αφορά τη χρήση των ε, πόρων ε, για την ανάπτυξη. Και θα ήθελα επίσης να επιμείνω στο θέμα του, της εμπορίας των ανθρωπίνων όντων. Εμείς επιμείναμε στην ανάγκη να δούμε το θέμα αυτό και ενδεχομένως όλες τις ε, πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να ληφθούν και τις επιχειρήσεις, για παράδειγμα Σοφία που, Σόφια που είναι, δεν, είναι, δεν θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική εάν δεν συμπεριλάβουμε το θέμα αυτό και θα πρέπει να συνεργαστούν όλες οι χώρες εδώ και στο πλαίσιο της συζήτησης για την απελευθέρωση των θεωρήσεων εισόδου με τις, ε, και να υποχρώσουμε τις χώρες εταίρους μας πραγματικά να εγκύψουν στο θέμα αυτό και με αυτό εννοώ συγκεκριμένα την ε, Τουρκία. Η ΛΥΜΠΕ, αυτό ανφέρεται στην έκθεση, αλλά νομίζω ότι είναι ιδιαίτερο σημαντικό να επιμείνουμε εδώ, επιμένει στην ανάγκη να μην εξαρτηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια από άλλες ε, πολιτικές γιατί αυτό αντιβαίνει στην ανάγκη να καταπολεμήσουμε τις αιτίες της μετανάστευσης που συνήθως είναι οικονομικές και κοινωνικές. Άρα λοιπόν η ανάπτυξη είναι α, απαραίτητο εργαλείο και δεν μπορούμε να το βάλουμε στην άκρη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόπες. <clears throat> Eh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να σας συγχαρώ για την εκλογή σας ως ε, Πρόεδρο της Επιτροπής και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο συνεισηγητές και τον κύριο Διαθεμέρα και την Έλενα Βαλενθιάνου για τα όσα έκαναν για να φτάσουμε μέχρι εδώ ε, με συμβαστικές προτάσεις με μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση που απασχολεί και την ε, πολιτική και δημόσια συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια πλήρη έκθεση που θεωρώ ότι αντιμετωπίζει με ευφυή τρόπο το θέμα της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δυνατότητα μετανάστευσης, ε, κυκλοφορίας, το νόμιμο έλεγχο αλλά και την νόμιμη δυνατότητα εισόδου και από μια ανθρωπιστική προπτική, δηλαδή ε, υποστηρίζοντας και τις αξίες που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να προσθέσω κάποια στοιχεία τα οποία ακούστηκαν βέβαια και από τις προηγούμενες παρεμβάσεις. Καταρχάς, ε, επειδή ε, δεν πρέπει να υπάρχουν παραδείγματα και συνέχεια των συμφωνιών ε, που έγιναν με την Τουρκία ε, και γιατί αυτό, διότι καταρχάς ε, δεν είναι στην ε, κοινοτική λογική και στον έλεγχο που πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συμφωνία με την Τουρκία δεν γνωρίζουμε καν τι νομική υπόσταση διαθέτει για παράδειγμα. Δεν υπάρχει διαβούλευση, δεν υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει συμμετοχή των διαφόρων θεσμικών οργάνων και της κοινωνίας των πολιτών. Και δεύτερον, διότι ε, τρόπον την να έχει και συνέπειες για τους ετούντε άσυλο. Και αυτό ε, δεν ε, πρέπει να το παραβλέπουμε. Για την περίπτωση της συμφωνίας με το Αφγανιστάν θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι είναι και η πλειοψηφία των όσων ήρθαν το 2016 και ε, γιατί θέτουν επιτάπητο τη δυνατότητα μαζικών επιστροφών και αυτό ε, απαγορεύεται και από το Διεθνές Δίκαιο και μπορεί ε, να γίνονται επιστροφές μόνο ε, συγκεκριμένων ατόμων όταν υπάρχει συμφωνία. Πρόκειται για τρία σημαντικά στοιχεία στις δύο αυτές τις συμφωνίες Τουρκία, με την Τουρκία και το Αφγανιστάν που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη στο μέλλον. Δεύτερον, θα ήθελα να σταθώ και στη γενικότερη προοπτική που έχει έκθεση για το πόσο σημαντικές θα είναι οι ε, μετατοπίσεις ανθρώπων, όχι μόνο η μετανάστευση, τα επόμενα χρόνια. Καρπός φυσικά της ανισότητας ευκαιριών και της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης που επικρατεί, αλλά όχι μόνο αυτό. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κριτήριο που έχουμε στη διάθεσή μας, ε, μετανάστευση και ε, ε, μετακινήσεις ε, για οικολογικούς λόγους που είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει να διαφαίνεται. Η Ευρώπη λόγω γεωγραφικής θέσης θα πρέπει να το αντιμετωπίσει και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια διότι υπάρχει και πολύ μεγάλη βία στη Μέση Ανατολή ε, και στη Βόρεια Αφρική. Και για να ολοκληρώσω τώρα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτά τα οποία βιώσαμε τα τελευταία χρόνια και αυτές οι μαζικές μετακινήσεις είναι και ένδειξη της αποτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική. Εδώ και ε, ε, λίγο καιρό συζητούσαμε το πόσο σημαντική είναι η εξωτερική μας πολιτική και το πώς θα μπορούσαμε να προσδώσουμε ασφάλεια στη γύρω περιοχή. Ε, το λέγαμε αυτό πριν από 10 χρόνια, έτσι, ε, πολιτική γειτονίας, η οποία πολιτική στην πραγματικότητα είναι εξωτερική πολιτική και κανονικά θα έπρεπε να οδηγήσει σε σταθερότητα, σε ανθρώπινα δικαιώματα στη γείτονα περιοχή μας. Αυτή τη στιγμή όμως είναι πολύ δύσκολο να παραβλέψουμε τα όσα συμβαίνουν και φυσικά θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την εξωτερική μας πολιτική λαμβάνοντας υπόψη και με τα όσα συνέβησαν στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή με εκατομμύρια ανθρώπους δυστυχισμένους. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο, κύριο ο κύριος Βάγκελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά στη νέα θέση που αναλαμβάνετε και είμαι σίγουρος ότι θα συνεργαστούμε πολύ καλά μαζί. Θα μιλήσω σλοβενικά. Poročili, o katerih se pogovarjamo, je sta dokaz zavesti, da imamo opraviti s problemom. Thank you. Ευχαριστώ. Πρόκειται εδώ για ένα πρόβλημα το οποίο έχει μεγάλη διάρκεια, θα έχει μεγάλη διάρκεια και θα πρέπει να επιλέξουμε μια προσέγγιση η οποία θα είναι πιο ενεργητική και η οποία θα αντιλαμβάνεται διαφορετικά τον κόσμο. Ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε μια νέα συγκυρία θα ήθελα να τονίσω ότι όλα τα προβλήματα τα οποία συνδέονται με τη μετανάστευση ε, θα πρέπει ε, να, ειδωθούν, να, τα προσεγγίσουμε συνολικά ε, σε ένα συνολικό πλαίσιο και να δούμε την, τις αιτιακές σχέσεις μεταξύ τους θα πρέπει να προσπαθήσουμε για μια ειρηνική διευθέτηση όλων αυτών των προβλημάτων. Γιατί μια πολιτική η οποία έχει νομιμοποιήσει την ε, βία ε, την, ε, και, την, κατάκτηση σχετίζεται ακριβώς με τις μεταναστευτικές ροές εκατομμυρίων ανθρώπων. Ίσως ακούσατε κάποια αποθαρρυντικά μηνύματα από την Ουάσιγκτον σε μια χιονοστιβάδα ειδήσεων οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα χαροποιές. Αυτό μας υποχρεώνει σε μια συνεργασία μεταξύ των χωρών και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μια συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών, των Υπουργείων Εξωτερικών, τα οποία είναι αρμόδια για, τα, για την ασφάλεια των μεταναστευτικών ροών. Αυτό στο παρελθόν ε, δεν έγινε με έναν ικανοποιητικό τρόπο και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι εμείς χρειαζόμαστε και την... Ε, ε, θα πρέπει μάλλον να παράσχουμε μεγαλύτερη βοήθεια προς τις χώρες που επιβαρύνονται ιδιαίτερα με τη μετανάστευση ε, τα τις χώρες της πρώην Βαλκανικής Οδού, της Μακεδονίας λέει ο μιλητής, αλλά και η Ορδανία και Λίβανο. Και δεν θα πρέπει εδώ να αρκεστούμε, να βλέπουμε εικόνες στην τηλεόραση για τα όσα υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, μια συνάδελφος είπε ότι και οι πρόσφυγες και οι ετούντες άσυλο και οι μετανάστες έχουν δικαιώματα τα οποία εδράσουν στο διεθνές δίκαιο και στα ανθρωπιστικά δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν να τους αφαιρέσουμε αυτά τα δικαιώματα γιατί στην περίπτωση αυτή θα αποποιηθούμε τα βασικά δικαιώματα του πολιτισμού μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. κυρία Σαφάουζερ έχει το λόγο. Ο κύριος Σαφάουζερ, συγγνώμη. Και εγώ θα ήθελα παρότι γίνεται σπάνιο αυτό να σας συγχαρώ Ελπίζω ως ε, πρόεδρος ε, θα ε, αποδεχθείτε αυτή την πραγματικότητα, τη νέα στις πολιτείες και απ' την άλλη θα αποδεχθείτε και το γεγονός ότι αυτό που συχνά αποκαλείται λαϊκισμός τελικά είναι μόνο ο δρόμος που ακολουθούν αυτοί που έχουν πληγεί από την παγκοσμιοποίηση και οι οποίοι δεν θέλουν να καταστραφούν. Και ότι αυτός ε, ο δρόμος ε, ε, αντιπροσωπεύει στη χώρα μου τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι λοιπόν ο δρόμος των λαών και οι λαοί αυτή τη στιγμή ξυπνούν. Σε ό,τι αφορά αυτή την έκθεση, θα ήθελα αρχικά να πω τα θετικά. Το θετικό, ας πούμε, είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η μετανάστευση ε, θα κλείσει και θα τελειώσει μόνο με ένα σχέδιο Marshall για την ανάπτυξη. Ε, και εγώ είμαι υπέρ ε, του ελέγχου των συνόρων μας σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, αλλά αυτή θα είναι μάταιη αν δεν εγκαθιδρύσουμε και στην Αφρική αλλά και αλλού ένα πραγματικό πρόγραμμα της ασφάλειας και της ανάπτυξης. Όμως θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η φιλοδοξία που έχουν οι λαοί είναι να μείνουν στην πατρίδα τους. Τι, το τι κάνουν η ελίτ τώρα είναι ε, να οδηγούν στη φτωχοποίηση όλες αυτές τις χώρες και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε ε, ο κόσμος να μπορεί να ευημερεί και να προοδεύει στην πατρίδα του. Αυτό σημαίνει ότι θα σταματήσουμε ε, αυτές τις συνεχείς επεμβάσεις και παρεμβάσεις που αποσταθεροποιούν τον, τις διάφορες περιοχές του κόσμου και περιφέρειες, Ιράκ, Λιβύη, η Συρία γιατί όλα αυτά δημιουργούν ε, καταστάσεις που εμείς οι ίδιοι έχουμε προκαλέσει και δεν είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε χωρίς ένα πραγματικό ε, πρόγραμμα ασφάλειας και ανάπτυξης ε, που θα οδηγήσει αυτό το νέο σχέδιο Marshall, αυτό το New Deal για τον κόσμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαχείριση και τον έλεγχο των συνόρων, αφήστε την προσοχή σα ε, στο γεγονό ότι η Μεγάλη Βρετανία προτίμησε ένα σκληρό ε, Brexit, μια σκληρή έξοδο, για να έχει τον έλεγχο των συνόρων τη. Γιατί αυτό ο έλεγχο συνόρων αποτελεί θεμελιώδε δικαίωμα των λαών. Θα πρέπει να το κατανοήσετε. Αφήστε επίση την προσοχή σα στο γεγονό ότι για μα η Γαλλία είναι κάτι το αδιαπραγμάτευτο ε, σε ό,τι αφορά τις ε, κινήσεις μας. Όμως αυτό είναι πολύ ευρύτερο. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη αυτή τη φιλοδοξία ε, των λαών. Δεν μπορείτε να την αγνοείτε και να την αρνείστε. Ένα δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να φέρω είναι η δικαιοσύνη. Όταν στα προάστια όπου έχουμε το μεγαλύτερο μέρος της μετανάστευσης, το 50% του πληθυσμού είναι άνεργο και όταν έχουμε ακόμα μεγαλύτερη μετανάστευση μετά, είναι η πρώτα και κύρια αδικία απέναντι ε, στους ε, μετανάστες που ήδη βρίσκονται στη χώρα μας και δεν βρίσκουν δουλειά ή που ακόμα και στη δεύτερη γενιά δεν καταφέρουν ε, να ενταχθούν στην κοινωνία μας. Υπάρχουν τέτοιοι που μας ψηφίζουν κιόλα. Σας προσκαλώ να αρθείτε στα δύσκολα προάστια στο Παρίσι. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που μας ψηφίζουν γιατί υπάρχει πρόβλημα δικαιοσύνης. Δεν ε, μπορούμε να αγνοούμε αυτές τις δύο πραγματικότητες. Ελπίζω η έκθεσή σας αρχικά να έχει τη φιλοδοξία για ένα πραγματικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Η έκθεσή σας να λαμβάνει υπόψη αυτό το πρόβλημα της δικαιοσύνης και να στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που έχει την ε, εμπειρία ε, στον τομέα της ανάπτυξης για πάνω από 20 χρόνια σε ό,τι αφορά τα ad hoc κονδύλια και μέσα που είναι απαραίτητα για να είμαστε αποτελεσματικοί και γρήγοροι. Γιατί αν ακολουθήσουμε τις συνήθεις διαδικασίες, γνωρίζω τι συμβαίνει για, παράδειγμα στην Υποσαχάρη Αφρική, όταν πάνε να υλοποιηθούν τα προγράμματα, ε, θα έχει ήδη περάσει ο ΑΕΣΙΣ και τα τεράστια μεταναστευτικά κύματα. Χρειαζόμαστε κατεπίγουσα δράσεις και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναλάβουμε ταχύτατα αυτή τη δράση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Σαφάζε. Επόμενος ομιλητής, Σκιώδη από την Επιτροπή ΔΕΒΕ, κύριο Γκερέρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ορισμένες φορές ε, οι μακροσκελείς παρεμβάσεις είναι πολύ καλές διότι ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Και νομίζω ότι η τελευταία παρέμβαση εξηγεί σαφέστατα για ποιο λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προχωρήσει με αυτή την έκθεση ε, επικεντρωνόμενοι ακριβώς ε, ε, σε αυτό το οποίο επιθυμεί η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επαναλάβαμε πάρα πολλές φορές την Επιτροπή Ανάπτυξης και ε, σήμερα και εγώ ως και όδης εισηγητής θα ήθελα να εκφράσω τη στήριξή μου στην εισηγήτρια της Επιτροπής Ανάπτυξης, αλλά, συγγνώμη, στον εισηγητή της Επιτροπής Ανάπτυξης, αλλά και στην εισηγήτρια της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που πιστεύω ότι έκαναν μια εξαιρετική δουλειά και πρέπει απαραίτητος να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία με ένα πραγματικό συμβιβασμό που θα τονίσει τα βασικά στοιχεία που θέλουμε να ε, τονίσουμε σε αυτή την έκθεση. Πρέπει να επαναλάβω ότι αυτό δεν ήταν μόνο στην Επιτροπή Ανάπτυξη, αλλά στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι θέμα που απασχολεί όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, συνάδει και με αυτά τα οποία εγκρίθηκαν στη Νέα Υόρκη και ε, επανειλημμένω. Ε, ε, επανάλαβε το Διεθνές Γραφείο Μετανάστευσης, διάφορες διεθνείς οργανώσεις, τα Ηνωμένα Έθνη για τους, για τους πρόσφυγες κλπ. Πιστεύω ότι στην έκθεση αυτή πρέπει να επισημάνουμε κάποια στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι η απάντηση σε αυτή την πραγματικότητα, που δεν είναι μια μεταβατική πραγματικότητα, αλλά ε, ένας οδικός χάρτης ο οποίος θα συμβιώσει και με εμά και με τον υπόλοιπο κόσμο για πάρα πολύ καιρό, για δεκαετίες ίσως, θα πρέπει να αποτελεί μια ε, μακροπρόθεσμη απάντηση. Δεν είναι απλώς η άμεση σπασμωδική αντίδραση σε συνέπεια κάποιας ε, συγκυριακής κρίσης ή μιας μαζικής αύξησης για ένα σύντομο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου και σε αυτή την περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα ε, με το βλέμμα στον ορίζοντα. Πρέπει λοιπόν να προσφέρουμε βιώσιμες Λύση η ανύψωση ενός τείχους δεν είναι βιώσιμη ε, λύση, είναι το εντελώς αντίθετο. Είναι μία λύση απαράδεκτη από πλευράς ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, καθόλου αποτελεσματική όσον αφορά το ρεύμα αυτών των ανθρώπων που ανέκαθεν κινούνταν στην ιστορία και θα συνεχίσουν να κινούνται και στο μέλλον. Δεύτερον, πιστεύω ότι η επιλογή να μην εγκαταλείψουμε αυτές τις χώρες οι οποίες αναλαμβάνουν το ουσιαστικό άχθος αυτών των μετακινήσεων είναι τόσο ηθική υποχρέωση, αλλά και στρατηγική πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ηθική υποχρέωση, διότι είναι ανήθικο να υπάρχουν χώρες οι οποίες υποδέχονται ένα πάρα πολύ αυξημένο ποσοστό ε, προσφύγων, για παράδειγμα τις περιπτώσεις του Λιβάνου ή της Ιορδανίας, και εμείς να έχουμε μια κρίση ε, την οποία κατά τα φαινόμενα δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όταν έχουμε απλώς μόνο το 0,5% του πληθυσμού, μας, ε, του πληθυσμού μας σε αντιστοιχεία προσφύγων που έφτασαν στην αποκαλούμενη αυτή κρίση. Και ε, δεν είναι βιώσιμο και από ηθικής και από στρατηγικής σκοπιάς, διότι Μόνο αν αυτές οι χώρες μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάλληλη διαχείριση αυτών των μεταναστευτικών ροών και των προσφύγων, θα μπορέσουμε να ε, έχουμε ειρήνη στο περίγυρο και να μπορέσουμε να απαντήσουμε με γεωστρατηγική ισορροπία στην κατάσταση που αυτή τη στιγμή αποτελεί κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως σκιώδης εισηγητής θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι Υποστηρίζω κατ' ουσίαν αυτό το οποίο λέγεται στην έκθεση όσον αφορά την ε, ε, δημιουργία νόμιμων οδών για να αντιμετωπίσουμε την ε, μετανάστευση, τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες. Νομίζω ότι και από τις προηγούμενες παρεμβάσεις υπάρχουν αντίστοιχες σκέψεις και ε, μας ενδιαφέρουν και οι διεθνείς συμφωνίες που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως συμφωνίες συνεργασίας για την ανάπτυξη και επίσης υπάρχει και η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο στις χώρες αυτές ε, με τις οποίες συνεργαζόμαστε, αλλά κυρίως εντός των συνόρων μας, διότι τις τελευταίες εβδομάδες ε, ε, είδαμε και κλιματική κρίση η οποία ε, οδήγησε σε θάνατο προσφύγων και ε, χιλιάδες εξ αυτών υποχρεώθηκαν να ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες και αυτό είναι ε, κατάφορη απόπειρα κατά των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων. Και Επίσης, θεωρώ ότι ε, στην έκθεση αυτή θα πρέπει να υποστηρίξουμε και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να υποχρεώσουμε το Συμβούλιο, τα μέλη του Συμβουλίου, να εφαρμόσουν όλα εκείνα που εγκρίθηκαν ε, στη διάρκεια του τελευταίου έτους, ε, τα οποία στην πραγματικότητα είναι ανεφάρμοστα. Ε, τις συμφωνίες για τους πρόσφυγες, τις συμφωνίες της Βαλέτας, να χρησιμοποιηθούν ε, τα compacts αυτά για τη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών του κόσμου και ούτω καθεξής. Με ξενοφοβία, με φόβο, με απόρριψη δεν θα λύσουμε τίποτα. Δεν θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα, θα το λύσουμε με σεβασμό στις ανθρώπινες ζωές, με συνεργασία και με μια στρατηγική ε, εικόνα που θα πρέπει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο, ιδιαίτερα σε αυτόν τον κόσμο που αρχίζει να εγκαταλείπει πολιτικά ε, τις ευθύνες του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω τρεις ακόμα ομιλητές. Λίτς, Κούσο και Σλάιν. Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Αν όχι, ε, στη συνέχεια θα ολοκληρώσει η κυρία Μακάβαν τη συνεδρίασή μα. και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λίτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θερμά συγχαρητήρια στην ε, εκλογή σας ως Προέδρου της Επιτροπής. Θα ήθελα να αναφερθώ στο όσα είπε ο κύριο Σαφχάουζερ από το Front National Πράγματι ελπίζω κύριε Σαφχάζερ ότι θα αφυπνιστεί ο λαός και θα αντισταθεί στο λαϊκισμό τον οποίο αναφέρεται. Προσπαθείτε να πείτε ότι τα πράγματα μπορούν να λυθούν εθνικά. Αντίθετα, μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να επιληθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Χαίρομαι πολύ που αυτή η ενεργό συνεργασία μεταξύ των εισηγητών εδώ είχε σαν αποτέλεσμα ένα πολύ καλό κείμενο, γιατί πράγματι χρειαζόμαστε μια νόμιμη μεταναστευτική πολιτική. Εκκλησίες όπως η Ιταλική Σεν Γκουίντο ήδη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Το ζητούμενο είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι χρειάζονται ανθρωπιστική βίζα να μας κάνουν να σκεφτούμε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε όλη την ευθύνη, όλο το φορτίο στις χώρες της ε, Νοτιού Ευρώπης. Εγώ ε, υποστηρίζω όλα αυτά τα προγράμματα γαλλογερμανικής ε, συνεργασίας. Η διασύνδεση μεταξύ κλιματικής πολιτικής και μεταστατικής πολιτικής είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το 2015 είχαμε μια γνωμοδότηση για να δείξουμε ότι η κλιματική πολιτική και η μεταναστευτική πολιτική είναι αλληλένδετες. Και στο βαθμό αυτό το, ε, ε, η έκθεση αυτή έρχεται και πάλι στο επίκεντρο της προσοχής μας. Τώρα όσον αφορά τον ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο, το Africa Trans Fund, ε, το Ταμείο Εκτακτής Ανάγκης για την Αφρική. Θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο θα πρέπει να συνεχίσουμε τη βοήθεια με την μορφή αυτή, θα πρέπει να είμαστε πιο ενεργητικοί. Το ίδιο ισχύει και για τις ε, μεταναστευτικές συμφωνίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει εδώ να συμμετάσχει πιο ενεργά, ε, συνδιαμορφώνοντας τα οικονομικά αλλά και την εξωτερική πολιτική. Η αναπτυξιακή συνεργασία ε, μπορεί να καταπολεμήσει τι αιτίε τη μετανάστευση. Και εμεί ω Κοινοβούλιο θα πρέπει να δείξουμε ξεκάθαρα ότι ε, σεβόμαστε του αναπτυξιακούς στόχου του 2013. Εδώ χρειαζόμαστε βεβαίω περισσότερα κονδύλια, ούτω ώστε το κλιματικό πακέτο των Παρισίων να μπορέσει να εκπληρωθεί, να εφαρμοστεί. Και ελπίζω πραγματικά να βάλουμε αυτά ως προτεραιότητες της ε, Προεδρίας της ε, Μάλτας. Ε, θα πρέπει να κάνουμε πραγματικά εμβληματικές πρωτοβουλίες και νομίζω ότι η έκθεση αυτή μπορεί να λειτουργήσει σαν βάση. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κούζο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το είπα και προηγουμένως, αλλά θα ήθελα και πάλι να σας συγχαρώ για την εκλογή σας. Για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να πω συνοπτικά ότι η έκθεση περιλαμβάνει κάποια θετικά στοιχεία και αυτό βεβαίως είναι καλό. Μου άρεσε πάρα πολύ που επαναλαμβάνεται κάτι το οποίο μας αρέσει ιδιαίτερα, η διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών, διότι υπάρχει αυτή η διάκριση. Η ε, μετανάστες ε, βρίσκονται σε μια κατηγορία στην οποία η νομοθεσία και οι συμβάσεις ε, που ε, έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να την χάνουν μια ευνοϊκή μεταχείριση την οποία εμείς δεν τους προσφέρουμε και πρέπει να το επαναλάβουμε αυτό. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή εντυπωσιακών μετακινήσεων πληθυσμών σε σχέση με το παρελθόν όπως έλεγε και ο ΙΕ μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που είχαμε τις μεγαλύτερε μετακινήσει πληθυσμών. Αυτό το οποίο δεν αναφέρεται όμως ε, στην έκθεση είναι το προπατορικό αμάρτημα και το προπατορικό αμάρτημα είναι οι παλαβή οι παλαβές παρεμβάσεις που έγιναν από το 2002 όταν έγινε μια προσπάθεια να ε, ανακατατάξουμε ε, στις ε, επιθυμίες κάποιων τρελών ανθρώπων τη Μέση Ανατολή. Ε, και ουσιαστικά ε, στα μέσα μαζικής ανημέρωσης δημοσιοποιήθηκε αυτός ο χάρτης που είχαν χαράξει κάποιοι στρατιωτικοί που οδήγησε σε ε, καταστροφή κάποιων ε, φυλών όπως, ή και χωρών όπως το Ιράκ, τη Λιβύη και τη Συρία. Εάν λοιπόν δεν ε, το έχουμε σαφώς αυτό στο μυαλό μας, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στη ρίζα του το πρόβλημα και να βοηθήσουμε αυτούς τους ε, πρόσφυγες, τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν βοηθάμε. Και το βλέπει όλος ο κόσμος. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ηθικά σφάλματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει επίσης ε, να υποστηρίξουμε το Λίβανο και την Ιορδανία. Ο Λίβανος είναι μια μικροσκοπική χώρα 7 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχει 2 εκατομμύρια προσφυγές προσφύγων. Όπως ε, ε, έκανε και στο παρελθόν η Συρία που υποδέχθηκε 2 εκατομμύρια Ιρακινούς. Ε, βρισκόμαστε λοιπόν σε μια συγκυρία στην οποία νομίζω συμφωνούμε τόσο εδώ όσον αφορά τα οικονομικά ζητήματα, όταν θα έπρεπε να καταπολεμήσουμε τις οικονομικές ασυμμετρίες, αλλά με ένα σαφές σχέδιο και να αντιμετωπίσουμε και ως ίσους τους γείτονές μας πρέπει να δράσουμε. Το βλέπουμε. Μετακινούνται οι πρόσφυγες λόγω του κρύου και ε, δεν υποστηρίζουμε χώρες όπως την Ελλάδα, ενώ κάποιες άλλες χώρες ε, δεν τηρούν συστηματικά τις συμφωνίες που έχουν γίνει για την ε, υποδοχή προσφύγων. Και ένα ακόμα σημείο με το οποίο διαφωνούμε είναι αυτή η πολιτική ασφάλειας και άμυνας και η πολιτική του ΝΑΤΟ για τα όσα γίνονται στη Λιβύα. Θα πρέπει να δούμε την χάρτα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε την ανθρωπιστική δυστυχία, ε, κάτι το οποίο δεν συνάδει και με το διεθνές δίκαιο. Ε, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε αυτό που έκανε η επιχείρηση Mare Nostrum που έσωσε 750.000 πρόσφυγες, κάτι το οποίο δεν κάνουμε εμείς γιατί βάζουμε ε, στην κορυφή της πυραμίδας τη στρατιωτικοποίηση και το γεγονός ότι δεν τηρούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, η κυρία Σλάιν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, δύο εισηγητές ε, για τη δουλειά που έχουν κάνει για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Πρέπει να πω ότι είμαι αρκετά επιφυλακτική ω προς την ε, τάση που ακολουθούμε σε ό,τι αφορά την μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική. Μετά την συμφωνία με την Τουρκία και την ε, πρώτη συμφωνία πλαίσιο με κάποιες αφρικανικές χώρες και μετά την πρόταση για την αναδιατύπωση του κοινού ε, μεταναστευτικού μάλλον συστήματος ασύλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε ότι υπάρχει ε, μία τάση να μεταθέτουμε μακριά από εμάς το πρόβλημα, μακριά από τα σύνορά μας, να μην το βλέπουμε, να μην μας απασχολεί και ε, να μην χρειάζεται να λαμβάνουμε δράση να βοηθούμε. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα συνοχή, συνάδελφοι, γιατί το Σεπτέμβριο ήμουνα στη Νέα Υόρκη, όταν για πρώτη ε, φορά συζητούσαμε το θέμα του μεταναστευτικού και προσφυγικού στην πρώτη λοιπόν Σύνοδο Κορυφή για αυτό το ζήτημα. Ε, και διοργανώθηκε αυτή η Σύνοδο Κορυφή με γνώμονα το γεγονό ότι το 86% όλων των εκτοπιστέντων στον κόσμο του υποδέχονται ουσιαστικά αναπτυσσόμενε χώρε. Επομένω, δεν είναι ευρωπαϊκό ζήτημα, είναι παγκόσμιο το θέμα τη ευθύνη. Αλλά πώ μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι όταν γενικά ζητούμε την, τον καλύτερο καταμερισμό της ευθύνη και δεν καταφέρουμε να το κάνουμε εμείς στο σπίτι μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπετε εικόνες των όσων συμβαίνουν στη Σερβία, στην Ελλάδα είναι προφανές. Δεν χρειάζεται ο συνάδελφος από το Front National να μας πει ότι είναι ε, αυτή, η κατάσταση και δεν μπορεί να συνεχιστεί. βεβαίω και είναι. Το 80% των αιτήσεων το διαχειρίζονται ένας πολύ μικρός αριθμός χωρών. Όμως πού είναι η αλληλεγγύη, πού είναι ε, ο ίσως καταμερισμός ε, των ευθυνών. Δεν είναι κάτι το οποίο εγώ ε, επινοώ. Ήδη υπάρχει στις συνθήκες μας το άρθρο 80 και 78. Γιατί μιλάμε λοιπόν εδώ τελικά. Ο συνάδελφος του Νασιονάλη είπε ότι υπάρχει πρόβλημα δικαιοσύνης. Όμως, δικαιοσύνη, κατά τη γνώμη μου, είναι μία έννοια αδιαχώριστα από τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι όταν ζητεί κανεί ε, διεθνή προστασία, αυτό είναι θεμελιώδη δικαίωμα και πρέπει να το, το χορηγήσουμε. Αν θέλουμε να ξεχάσουμε και τη νομική αλλά και ηθική ευθύνη που έχουμε ε, ενώπιον αυτών των ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τους πολέμους και τις ε, καθελογής διώξεις. Ναι, οποιοδήποτε μπορεί να βγει στον δρόμο και να δώσει την εικόνα ότι υπάρχει μία ε, εισβολή στην Ευρώπη. Τα προάστια στα οποία αναφερθήκατε αδελφά, όπου ε, υπάρχει έλλειψη οποιασδήποτε προοπτικής ε, θέσης εργασίας, κοινωνικής δικαιοσύνη που θα τους βοηθούσε να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά του προβλήματα. Δεν εκπλήστε κανεί που φοβούνται λοιπόν, Όμω είναι πολύ ανεύθυνο να εκμεταλλευόμαστε αυτό το φόβο όπως κάνουν κάποια κόμματα και να χρησιμοποιούμε τους μετανάστες ως αποδιοπομπαίους ε, τράγους ε, για την αδυναμία του πολιτικού μας συστήματος να τους στηρίξουν έναντι της ε, ανεργίας. Ποιος ευθύνεται λοιπόν γι' αυτό οι μετανάστες, μα είμαστε σοβαροί. Πρέπει επίσης να, να μην δημιουργούμε και μία ψευδή εικόνα της ε, κατάστασης, της πραγματικότητας, που είναι πραγματικά σκληρή. Θέλετε να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους στη χώρα τους. Ας σταματήσουμε λοιπόν τη φορολογική πολιτική ευρωπαϊκών εταιριών που χρησιμοποιούν ε, ως φορολογικούς παραδείσους ολόκληρες ε, αφρικανικές χώρες. Τα τελευταία 50 χρόνια η Αφρικανική Ένωση λέει ότι οι αφρικανικές χώρες έχουν χάσει περίπου 1-3 δολάρια εξαιτία τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή των δικών μα επιχειρήσεων, όχι των δικών του. Είναι περίπου το ποσό που λαμβάνουν σε αναπτυξιακή βοήθεια. Επομένω, με το ένα χέρι παίρνουμε αυτό που δίνουμε με το άλλο χέρι. Α σταματήσουμε λοιπόν αυτές τις εμπορικές συμφωνίε που έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε αυτές τις χώρες. Α σταματήσουμε να εκμεταλλευόμαστε τους φυσικού τους πόρου. Αν συνάδελφοι λοιπόν ψάχνετε να βρείτε τους λόγους για τους οποίους αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στη χώρα σας, μάλλον θα τους βρείτε πολύ πιο κοντά από ό,τι πιστεύατε. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο η Συμπροέδρος κυρία Μακάβων για το κλείσιμο. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα και εγώ ε, να συμφωνήσω με όλους τους υπόλοιπους που σας συνεχάρισαν ε, κύριε Μακάλιστερ για την εκλογή σας ως Προέδρου στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, ευχαριστώ τους δύο συνεισηγητές για τη δουλειά που έχουν κάνει, ε, για την επίτευξη συμβαστικών λύσεων. Βλέπω ότι υπάρχουν 37 συμβαστικές τροπολογίες, οπότε η ψηφοφορία την επόμενη φορά θα είναι πολύ πιο εύκολη μία τελευταία παρατήρηση. Εντάξει, υπήρξαν πολλέ τροπολογίε, μεγάλη έκθεση, αλλά πρέπει να είναι και σαφέ το μήνυμα του Κοινοβουλίου την επόμενη εβδομάδα. Να ε, τονισουμε τεσσερα τέσσερα-πέντε σημεία για να ξέρουν και ξέρει και το ευρύ κοινό περί τίνος πρόκειται. Γιατί ε, για πρώτη φορά αναλαμβάνουμε όλοι μαζί αυτό το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής. Πιο παλιά το ζήτημα το μεταναστευτικό αφορούσε περισσότερο τη ΛΥΒΕ και επιμέρους επιτροπές. Αλλά είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό. Την επόμενη Τρίτη λοιπόν, 31η Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε στις 3 το απόγευμα 4 την έκθεση αυτή. Αλλά θα ενημερωθείτε και για την επόμενη κοινή επιτροπή για αυτή τη σημαντική ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Επιστρέφω το λόγο στον ε, κύριο Μακάλιστερ. Ευχαριστώ πολύ για τη σύνοψη. Υπό τα διάφορα. Υπάρχει κάτι. Όχι. Ας κλείσουμε λοιπόν εδώ την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας με την Επιτροπή ε, Ανάπτυξης ε, και ευχόμαστε καλή συνέχεια στους συναδέλφους. Είναι 10.30. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε στην τακτική μας συνεδρίαση. Ας περάσουμε στο σημείο 10 ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη σημερινή κατάσταση και τις αυξανόμενες εντάσεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα μας απασχολήσει ένα ζήτημα το οποίο έχει αναλάβει αρχικά ο κύριος Ιβο Βάγκελ, συνάδελφός μας από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, και πρότεινε να συζητήσουμε τις πρόσφατες εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια στην Επιτροπή μας. Και νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα εφόσον ε, ε, παρατηρούνται αυξανόμενες εντάσεις ε, στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες. Και πολύ συχνά έχουμε αναφέρει στην Επιτροπή μας ότι αυτή η περιφέρεια βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης και περιτριγυρίζεται από ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και οι εξελίξεις ε, στην περιοχή αυτή έχουν άμεσο αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω σε περίοδους ε, κρίσης και αναταραχής. Θα πρέπει να θεωρούνται περιοχές ύψή ε, της προτεραιότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προκλήσει που αφορούν και πλήττουν σχεδόν όλες αυτές τις χώρες στην περιοχή αφορούν την ελλειπή συμφιλίωση, τις, τις και την έθραυστη ειρήνη που υπάρχει, τον κίνδυνο της ε, Ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης, την αυξανόμενη επιρροή της Ρωσίας, ε, ελλειπή πολιτικό διάλογο ε, μεταξύ άλλων. Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις προσθέτουν και επιτείνουν αυτές τις εντάσεις, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη αντιπαράθεση μεταξύ Σερβίας και Κωσοφοπεδίου για το ζήτημα με το τρένο, αλλά και στην πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας, μετά τις εκλογές, η αυξανόμενη εθνική πόλωση στη Βοσνία και Ζεγοβίνη, το υποτιθέμενο πραξικόπημα, η απόπειρα πραξικοπήματο στο Μαυροβούνιο την ημέρα των εκλογών και πιθανή ε, ρωσική εμπλοκή. Όλα αυτά δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να μα απασχολήσει και μας εδώ στο Κοινοβούλιο αυτό το σημαντικό ζήτημα και ευχαριστώ τον κύριο Βάγκελ που το έφτιαξε. Να δώσουμε πρώτα τον λόγο στους ε, συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον κύριο Πρέντα, συντονιστή από πλευράς ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, γνωρίζετε ότι συνδυάζεται η ποιότητα, συνδυάζεται η το, τον συντονισμό με την ιδιότητα του εισηγητού για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πολύ που έχουμε σήμερα μια συζήτηση για τα Δυτικά Βαλκάνια, για τις σχέσεις ε, που έχουμε με την ε, περιοχή αυτή. Και νομίζω ότι το ενδιαφέρον που έχουμε σήμερα για τις ε, εντάσεις που συνεχίζουν να σοβούν ε, στην περιοχή αυτή εξηγείται το ενδιαφέρον αυτό από δύο λόγους. Καταρχήν θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική κρίση της δημοκρατίας στις χώρες της περιοχής αυτής των Δυτικών Βαλκανίων το εκλογικό σώμα ε, συνεχίζει να ελκύεται από τις λεγόμενες εθνο, εθνικιστικές ε, πολιτικές και οι εθνοτικές ε, διαρρέσεις κινητοποιούνται προκειμένου να προσελκυστούν ψήφοι. Οι εκλογικοί περίοδοι δείχνουν ότι ο εθνικισμός κυριαρχεί από την άλλη υπάρχει η αυξανόμενη περιοχή της Ρωσίας, επιρροή συγγνώμη της Ρωσίας στην περιοχή αυτή και στη Ρωσία ε, το εθνιστικό στοιχείο της ε, πολιτικής ε, έχει επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιρροή της Ρωσίας είναι τόσο στη Βοσνία όσο και στην Ρεπούμπλικα Σέρψκα πριν από μερικές ε, μέρες ε, διεξήχθη Συγγνώμη, συνάδελφε, κύριε Σαφχάουζερ, μπορείτε να συνεχίσετε έξω τη συζητήσεις σας. Κύριε Πρέντα, παρακαλώ. Ναι, έλεγα λίγες μέρες πριν από το δημοψήφισμα στη Ρεπούμπλικα Σέρψκα, εδώ και μερικούς ε, μήνες, υπήρξε ξεκάθαρη υποστήριξη εκ μέρους της Μόσχας για αυτή την ε, ε, πράξη που είναι αντισυνταγματική. Και θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν και κάποια θετικά ε, σημεία στη Βοσνία Ριζαγωνίνη. Χθες ο πρόεδρος ήταν στο, είχε μετέβει στο Βελιγράδι για έναν διάλογο με τους γείτονές του. Αυτό είναι θετικό. Όμως παρόλο που υπάρχει μεγάλη σύγχυση εδώ και θα πάρα πολύ να πυροδοθεί μια έκρηξη στην περιοχή. Εδώ και 2014 ε, λέγεται ότι η διεύρυνση θα γίνει, θα αναβληθεί για αργότερα και από αυτό αποφελούνται οι, οι εχθροί της Ευρώπης, οι εχθροί του εξυγχρονισμού. Και στη δική μας ε, χώρα, σε εθνικό επίπεδο, ε, καμιά φορά βλέπουμε να ενθαρρύνονται οι αποκλήσεις αυτές προς ε, μη δημοκρατικές διαδικασίες στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέδα. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε φορά που συζητούμε ζητήματα των Βαλκανίων έχουμε ένα μακρύ κατάλογο μιλητών. Παρακαλώ λοιπόν να είστε ή δυνατόν σύντομοι ούτως ώστε να μπορέσουν όσο δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι να μιλήσουν. Επόμενο ο μιλητής, ο κύριος Πίτσολα από τους σοσιαλιστές. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερως ε, που εξετάζουμε σήμερα στην Επιτροπή μας αυτό το ζήτημα, γιατί πάντα με πολύ ανοιχτό πνεύμα εξετάζουμε την πολιτική κατάσταση και τις πολιτικές σχέσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και όπως έχουμε πει πολλάκις, τα Δυτικά Βαλκάνια όντως ε, τους αξίζει ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Ταυτόχρονα όμως πάντα ξεκάθαρα λέμε ότι τίνουμε μια χείρα βοηθείας ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως θα πρέπει αντίστοιχα χείρα να τίνουν και ε, τα Δυτικά Βαλκάνια και να αναλάβουν ε, την ευθύνη κάθε χρόνο να αποδεικνύουν ότι όντως έχει σημειωθεί πρόοδος η οποία μετράται με τη δυνατότητά τους να υιοθετούν ευρωπαϊκά πρότυπα πρώτα απ' όλα θα πρέπει να θεσπίσουν ε, σχέσεις συνεργασίας στην περιοχή τους. Μια περιφέρεια που μέχρι πρόσφατα ε, γνώρισε την καταστροφή εξαιτία του πολέμου και γι' αυτό δεν είναι εύκολο ε, να μετρήσουμε ακριβώς την πολιτική πρόοδο, γιατί πάντα μπορεί κανείς να κινήσει, να προβεί σε τέτοιες πολιτικές ενέργειες που να υπονομεύσουν τη σταθερότητα. Νομίζω ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν από δύο παράλληλε διαδικασίε. Πρώτον, ε, πώς κινούνται ε, αυτές οι χώρες ως προς, τις, ε, προς την ενταξιακή τους πορεία αλλά και πώς ε, λειτουργούν οι δυνάμεις που αντιτίθενται στην, ε, στο ευρωπαϊκό όραμα. Νομίζω ότι υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις και στο εσωτερικό των Δυτικών Βαλκανίων. Όμως ε, η πρόοδος αυτών των δυνάμεων μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις μεταξύ των χωρών. Αυτό βλέπουμε στην περίπτωση του τρένου αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιβραδύνει ακόμα περισσότερο την οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινα. Έχει σημειωθεί πρόοδος, η οποία όμως μπορεί να επανομευθεί από τις πρόσφατες εντάσεις. Οι χώρες ε, των Δυτικών ε, Βαλκανίων γνώρισαν μεγάλες δυσκολίες το 2015 και 2016 λόγω του μεταναστευτικού αλλά και των διαφορών εκλογικών αναμετρήσεων. Εκ πρώτης όψεως δεν έχει αλλάξει κάτι. σε ό,τι αφορά την ε, αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως προς αυτή την ε, περιοχή, σε αυτές τις χώρες όμως ε, υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια ε, τα οποία μπορούν να θέσουν ένα αμφιβόλο την ευρύτερη διαδικασία. Γι' αυτό και χαιρετίζω την συνάντηση που θα λάβει η χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες μεταξύ Κοσμοπεδίου και Σερβίας Γιατί και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση της Μακεδονίας, λέει ο ε, είναι έτσι η κατάσταση που μπορούν όλα πραγματικά ε, να ε, διακινδυνευτούν και να διακινδυνευτεί έτσι και η ευρωπαϊκή εξέλιξη. Ο κύριος Βάγκελ. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πάρω το λόγο γιατί το θέμα αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερος και είναι και εξαιρετικά επίκαιρο. Εγώ προέρχομαι από την περιοχή αυτή, όπου πραγματικά συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας ανησυχούν και για τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε εγκαίρως. γιατί έτσι όπως ε, ήταν οι εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή είδαμε ότι από μια μικρή σπίθα μπορεί να δημιουργηθεί μια μεγάλη ανάφλεξη, μια πυρκαγιά. Θα ήθελα να πω καταρχήν γιατί ανέλαβα την πρωτοβουλία για, την, ε, για να γίνει αυτή η συζήτηση. Στο Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή γίνεται η προετοιμασία μιας έκθεσης για την ε, πρόοδο των χωρών της Νοτιοανατολικής ε, Ευρώπης. Στις εισηγήσεις αυτές εγώ είμαι, είμαι για την Μακεδονία, λέει ο, ο μιλητής, και στην έκθεση αυτή ε, θεωρούμε δεδομένο ότι θα πρέπει να συνεχίσει, θα πρέπει να δοθεί μια συνέχεια στην επιθυμία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό δεν θα χρησιμεύσει μόνο στις ε, χώρες αυτές και στους λαούς αυτούς, αλλά και στη σταθεροποίηση αυτού του τμήματος της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Επίρου. Όλα, ε, όλες οι διαφωνίες που ενδεχομένω υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης μπορεί βεβαίως να αναχαιτήσει τη διαδικασία ένταξης και μπορεί να αποδυναμώσει την ε, βούληση για πολιτική υποστήριξη ε, των χωρών αυτών τους να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, την υποστήριξη υπέρ για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η διαδικασία θα μπορούσε να αναχαιτιστεί με τον τρόπο αυτό. Και η δική μου επιθυμία ήταν εδώ να μεριμνήσουμε έγκαιρα, ούτως ώστε να κερδίσουμε την ε, προσοχή της Ευρώπης για το θέμα αυτό. Στην πρώην χώρα δημοσιεύθηκε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Ο, ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7.30». Ε, και το βιβλίο αυτό επισημαίνει το γεγονός ότι όλοι, όλες οι σειράξεις και οι πόλεμοι στην περιοχή αυτή ξεκινούν με μια ρητορική μίσους. Και πολλά στοιχεία εδώ αναγνωρίζουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στοιχεία αυτής της ρητορικής του μίσους. Και δυστυχώς ακόμα και πολύ διακεκριμένοι εκπρόσωποι της πολιτικής συμμετείχαν σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Ε, έχω ορισμένες τέτοιες δηλώσεις ε, της ρητορικής μίσου, δεν πρόκειται να σας τη διαβάσω, αλλά η ανησυχία πραγματικά ε, ε, ιδιαίτερη μεγάλη ανησυχία ε, εκδηλώθηκε όταν ο πρόεδρος της ε, Σερβίας μίλησε, αναφέρθηκε μάλλον σε έναν επικείμενο πόλεμο στην περιοχή αυτή. Και υπήρξαν και πολλές άλλες τέτοιες δηλώσεις προς την κατεύθυνση αυτή που πραγματικά δίνουν λαβή σε σοβαρότατες ανησυχίες. Ευχαριστώ. Έχουμε 11 αγορητές στο κατάλογο, απλώς ενημερωτικά. Η κυρία Λούνατσεκ έχει το λόγο στη συνέχεια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση Και εγώ την περίμενα γιατί πραγματικά ανησυχώ ιδιαίτερα για τα όσα συνέβαιναν, όχι μόνο στη χώρα που γνωρίζω καλύτερα, διότι είμαι και εισηγήτρια για το Κωσυφοπαίδιο, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ Σερβίας Κωσυφοπαιδίου και άλλες χώρες όπως για παράδειγμα η Βοσνία Ριζογοβίνη, η Ρεπούμπλικα Σέρψκα, το Μαυροβούνιο κλπ. Αυτό ε, σημαίνει ότι και η ανησυχία που εξέφρασαν οι συνάδελφοι είναι ανησυχία την οποία συμμερίζομαι και εγώ. Εμείς λοιπόν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιδείξουμε πολύ μεγαλύτερο στένος ε, και το Κοινοβούλιο όμως αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να ζητήσουμε από όλες τις κυβερνήσεις αλλά επίσης ε, και από άλλους φορείς ε, στις έξι χώρες των Βαλκανίων να επικεντρωθούν στις ευρωπαϊκές αξίες, α το πω έτσι. Διότι ένα από τα στοιχεία που αποτελούν την ουσία της ε, διαδικασίας της διεύρυνσης και ένα από τα στοιχεία που αποτελούν την ουσία της ε, δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ξεπεράσουμε τις εθνικιστικές απειλές, οι οποίες ε, τον τελευταίο αιώνα έφεραν στην Ευρώπη τους πιο βίαιους ε, πολέμους και τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα. Αυτό προϋποθέτει καλές γειτονικές σχέσεις και με ανθρώπους που υπήρξαν εχθροί και που ε, πολέμησαν ο ένας τον άλλον πριν από λίγες δεκαετίες και μόνον έχω την εντύπωση με όλα αυτά τα οποία ε, βιώνουμε τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες ε, και τώρα και με την εκλογή του κυρίου Τραμπ στις Ηνωμένε Πολιτείες ε, στηρίζονται πολλές φορές ακραίοι εθνικιστές που δεν θέλουν να δεχτούν ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαφορετική γλώσσα, πιστεύουν ίσως σε διαφορετική θρησκεία, αλλά που ήταν ε, γείτονες στην πρώην Ιουγκοσλαβία πριν από 30 χρόνια, δεν είναι παρά άνθρωποι. Και νομίζω ότι ορισμένε φορέ υποχρονόμαστε να συζητούμε αυτά τα βασικά στοιχεία. Άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν στη Ιουγκοσλαβία, που είναι τώρα εδώ μαζί μα, γνωρίζουν πώ έχει η κατάσταση. Εγώ γνωρίζω λόγω των επισκέψεων ε, που έκανα και δεν θέλω φυσικά να επανενωθεί η Ιουγκοσλαβία, μην με παρεξηγήσετε, αλλά θέλω αυτά τα ευρωπαϊκά ε, θέματα, όπω για παράδειγμα οι καλέ γειτονικέ σχέσει να ε, τα προωθήσουμε. το θέμα του τρένου, για παράδειγμα, που εστάλει από Σερβία στο Κωσυφοπαίδιο πριν από λίγες ημέρες ε, που έλεγε ότι το Κωσυφοπαίδιο είναι σερβικό και ε, μέσα ήταν εθνικιστές οι οποίοι έλεγαν αυτά τα οποία ε, πρεσβεύουν. Ε, και αυτά χρηματοδοτήθηκαν και από κυβερνήσεις. Ε, ε, χαίρομαι λοιπόν που σήμερα γίνεται ένας διάλογος στις Βρυξέλλες με το Κόσοβο και τη Σερβία να κάθονται δίπλα-δίπλα και να συζητούν. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε και να προωθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που επιθυμούν τις ευρωπαϊκές αξίες σε αυτές τις χώρες. Αυτό λοιπόν το οποίο με ενδιαφέρει σήμερα είναι να δούμε πώς μπορούμε εμεί ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πιέσουμε για μεγαλύτερη συνεργασία. Υπάρχει για παράδειγμα ε, το σχέδιο της ε, περιφερειακής συνεργασίας των νέων, ένα πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στις χώρες αυτές, στα πλαίσια της διαδικασίας του Βερολίνου. Χρειαζόμαστε περισσότερες τηλεοπτικές εκπομπές, βιβλία ιστορίας, τα οποία θα εξετάζουν πώς συνομιλούν οι γείτονε και δεν θα υποκινούν το, ε, το μίσος και θα προωθούν περισσότερο μίσος και βία. Διότι αυτό είναι οπισθοδρόμηση και όχι η πρόοδος. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Σαφχάουζερ. Ακούω αυτό που είπε η συνάδελφος Λούνατσεκ, να επικεντρωθούμε στις ευρωπαϊκές αξίες και διαρωτώ με κατά πόσον οι ευρωπαϊκές αξίες είναι αυτές οι οποίες μας οδήγησαν στον βορμαδισμό της Σερβίας για να θεμελιώσουμε τη δημοκρατία. Αυτές είναι οι ευρωπαϊκές αξίες. Και αναρωτιέμαι μήπως ευρωπαϊκές αξίες είναι αυτές οι οποίες μας εξώθησαν να αναγνωρίσουμε το κοσφοπέδιο, παρά το γεγονός ότι είναι μια χώρα η οποία δεν είναι αναγνωρισμένη σε διεθνές επίπεδο προς το παρόν από όλες τις ε, διεθνείς οργανώσεις και να κάνουμε ένα κράτος μαφίας κράτος. Είναι αυτές οι ευρωπαϊκές αξίες. Την ακούω να καταδικάζει τον εθνικισμό. Ο κύριος Μποστινάρ διακόπτη ως χώρα που δεν αναγνωρίζει το κοσφοπέδιο, το να συζητάτε για μια χώρα που είναι αναγνωρισμένη από το Ηνωμένα Έθνη δεν είναι κράτος, είναι απαράδεκτο. Και εσείς κύριε Πρόεδρε θα πρέπει να τον διακόψετε. Ο κύριος Μακάλιστερ. Κύριοι, κύριοι, συνάδελφοι, ε, είμαι συνηθισμένο στι δηλώσει του κ. Σαπχάιζερ. Ε, περίμενα να συνοψίσω στο τέλο τη δήλωσή του, διότι δεν θέλω να του δίνω και τόση προσοχή. Αγαπητέ συνάδελφοι, σα παρακαλώ σταματήστε να αποκαλείτε το κοσυφοπαίδιο με του όρου που χρησιμοποιήσατε. Είναι ε, απαράδεκτο και θα πρέπει όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε να την χάνουν του ίδιου σεβασμού. Ευχαριστώ. μπορείτε να συνεχίσετε τώρα, χωρίς να χρησιμοποιείτε τέτοιους χαρακτηρισμούς για το κοσμοπέδιο. Ε, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε, μπορώ να μιλήσω και ξύλινη γλώσσα, αλλά η αλήθεια δεν θα αλλάξει. Η αλήθεια είναι πολύ πιο ισχυρή και ακόμα και η αλήθεια της ευφυΐας ε, ε, κάποιων ε, ε, γερμανικών επιχειρήσεων και ότι κάνουν διάφορα δίκτυα. Και κάποια στιγμή όλα θα έρθουν στην επιφάνεια. Γνωρίζετε την ιστορία, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά η αλήθεια εξακολουθεί να υπάρχει. Εσείς καταδικάζετε τον εθνικισμό. Σαφώς και υπήρχε πρόβλημα εθνικισμού. Αλλά ε, να σας υπενθυμίσω την ε, ιστορία της Ευρώπης ε, όταν ε, μας επιτέθηκαν. Το 1914 και το 1918 δεν μας επιτέθηκε η Γαλλία. Το 1940 και 1941 δεν ήταν η Γαλλία αυτή η οποία επιτέθηκε. Και είναι αλήθεια ότι στη Γερμανογαλλική Συμμαχία θεμελιώσαμε την Ευρώπη. Αλλά δεν θα πρέπει να έχουν την ίδια ευθύνη όλες οι πλευρές. Δεν είναι στη χώρα μου η ευθύνη. Η χώρα μου είναι αυτή η οποία θεμελίωσε και θέλησε αυτή τη νέα συμφιλίωση μεταξύ Γερμανία και Γαλλία. Ναι, να καταδικάσετε τον εθνικισμό, αλλά όχι τον τυχαίο εθνικισμό. Τον εθνικισμό ο οποίο είναι πολεμοχαρή, ο οποίο οδηγεί σε πολέμου. Και να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι και όλες τι χώρες στο ίδιο καζάνι, να επανέλθω στη Γιουγκοσλαβία Υπήρχε μια τάση και στους Αψβούργους ε, ε, μετά από τη Ιουγκοσλαβία να γίνει μια ένωση και να υπάρχει μια ομοσπονδία. Και εμείς αυτό το εμποδίσαμε, θα πρέπει να το πούμε, πρέπει να επενθυμίσουμε την ιστορία. Ε, ποια ήταν η πρώτη χώρα η οποία αναγνώρισε και δεσμεύτηκε σε αυτήν όλη διαδικασία. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σωστοί. Επανέρχομαι στο θέμα του ποιος είναι σωστός. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε πάντα ε, λέμε ότι είναι καθήκον μας να σεβόμαστε τις μειονότητες. Αλλά μπορείτε να αντιληφθείτε ότι οι Σέρβοι στη Βοσνία Ζεβοβίνη ε, που ορισμένες φορές είναι και το 40% του πληθυσμού σε κάποιες περιοχές της Βοσνίας. Θα πρέπει λοιπόν να πείτε, διακόπτει ο Πρόεδρος, Τελείωσε ο χρόνο αγόρευσή σα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να σα ζητήσω να μην προεδρεύετε στον κύριο Μπροκ και να αφήνετε και την αντιπολίτευση να μιλάει. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαφχάιζερ, όλοι έχουν όλοι τον ίδιο χρόνο αγόρευση και το αυτό ισχύει και για εσά. Αυτό είναι το λογικό. Η κυρία Σουίτσα, η αντιπρόεδρό μα τώρα. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακάλιστερ. Συμφωνώ με τα όσα μας είπε η κυρία Λούνα Τσέκ. Επιθυμείτε διαφορετικούς μηχανισμούς, αποστολές, ανταλλαγές φοιτητών, καλά όλα αυτά. Αρκεί βέβαια και οι ηγέτες τους να ακολουθήσουν ε, την ίδια οδό. Εγώ θεωρώ ότι οι λαοί της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ε, και των Δυτικών Βαλκανίων είναι υπέρμαχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξακολουθούν να στηρίζουν την ένταξή τους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά πλειονότητα. Το πρόβλημα εδώ είναι η συμμόρφωση των ηγετών τους. Εγώ προέρχομαι από την Κροατία, από την ίδια δηλαδή περιφέρεια. Δεν θέλω λοιπόν ε, να διαλέξω μέρος, αλλά η αλήθεια είναι ότι η ευθυγράμμιση με τη Ρωσία δημιουργεί πολύ σημαντικά προβλήματα. Πρόβλημα υπάρχει και με την ε, ελευθερία του τύπου σε κάποιες αυτές τις χώρες. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εκφράσει τη βούλησή του να παρακολουθεί στενά τις πολιτικές εξελίξεις ε, σε αυτή την περιφέρεια, θα έχουμε περαιτέρω υπονόμευση της δημοκρατίας εκεί. Έχουμε λοιπόν αιτήσεις εκθέσεις προόδου, όμως αυτό δεν φτάνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι παρούσα στην περιοχή και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στη διατήρηση της σταθερότητας εκεί. Δεν μπορούμε λοιπόν να παραμελούμε ή να γνωρούμε αυτή την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Ε, ούτε να τη βγάλουμε από τον κατάλογο προτεραιοτήτων μα. Ο μοναδικό τρόπο διατήρηση τη σταθερότητα είναι η συνεχής παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό απεδείχθη ήδη στις περιπτώσει τη Σλοβενία και τη Κροατία, και ελπίζω ε, να βοηθήσουμε και άλλες ε, χώρες να ακολουθήσουν ε, τον ίδιο δρόμο. Το Brexit έχει γίνει κύριο θέμα συζήτησης και δυστυχώς ε, ελοχεύει ο κίνδυνο και οι εσωτερικέ μας συζητήσει ε, να ε, επικεντρώνονται μόνο σε αυτό το θέμα και έτσι να περιθωριοποιηθεί το ζήτημα των Δυτικών Βαλκανίων. Και νομίζω ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Μια πιθανή ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το βασικό κίνητρο για όλες αυτέ τι χώρε. Η εξελίξη των τελευταίων ημερών, λοιπόν, νομίζω ότι κυρίως ε, προκύπτει από, από εσωτερικέ αιτίε σε αυτέ τι χώρε. Ευχαριστώ τον κύριο Βάγκελ που ε, έθιξε αυτό το ζήτημα. Είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν νομίζω ότι θα κλιμακωθούν αυτές οι εντάσεις περαιτέρω. Όμω θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα στι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων και είναι ο μοναδικό τρόπο ε, να ευημερήσουν αυτέ οι χώρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φαγιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον ε, την περιοχή. Ε, με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα όσα συμβαίνουν εκεί και χαίρομαι που έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα ανάβουν τα αίματα και έτσι πρέπει, γιατί δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς με τα όσα συμβαίνουν. Γιατί εγώ έρχομαι σε επαφή με νέους που βλέπω ότι θυμώνουν, ε, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, γιατί βλέπουν συνεχώς ε, αυξανόμενο εθνικισμό και μετανάστευση προς το εξωτερικό των νέων και ε, υψηλά καταρτισμένων. Πολλέ φορέ ε, οι ίδιοι λαοί μα λένε ότι τα πηγαίνουν καλά μεταξύ του, αλλά οι πολιτικοί είναι αυτοί που προσπαθούν να μα χωρίσουν. Γι' αυτό και δράτω την ευκαιρία για να αναφέρω ότι θα πρέπει όλοι να απέχουν από τους εθνικιστικούς αυτούς λόγους. Είναι πολύ ε, επικίνδυνος αυτός ο δρόμος γιατί ξυπνούν ε, μνήμες πολέμου καταστροφών και αβεβαιότητας και δεν θα πρέπει να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Δυστυχώς δεν μπορώ ε, να μην πάρω το λόγο σε σχέση με αυτό το περιστατικό με το τρένο, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει ε, μια ευκαιρία ε, συμφιλίωση των δύο λαών, περαιτέρω συμφιλίωσης και ε, ουσιαστικά προκάλεσε ε, ένα έναυσμα λαϊκιστικών και εθνικιστικών ανταλλαγών πυρών εντό εισαγωγικών μεταξύ των δύο χωρών είναι απαράδεκτο. Το ίδιο έχει γίνει και με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, με την Κροατία, σε κάποιε περιπτώσει και στη Μακεδονία πρόσφατα. ο Γκρουεύτσκι επιτέθηκε σε μη κυβερνητικέ οργανώσει ότι ενεργούν κατά των συμφερόντων τη χώρα του. Όλο αυτό είναι πολύ δυσάρεστο, οδηγεί τους νέους στη μετανάστευση, δεν βοηθά στη συμφιλίωση. Και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που συνεχίζεται ο διάλογο σήμερα στις Βρυξέλλες μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας. Έχει έρθει η ώρα για ανοιχτό διάλογο ε, και να σταματήσει η επικίνδυνη αυτή ρητορική ε, στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαγιόν. Έχουμε ακόμα 10 ομιλητές. Θα κλείσουμε τώρα τον κατάλογο ομιλητών. Και τώρα θα πρέπει να περιορίσουμε τον χρόνο αγόρευση στα δύο λεπτά. Ο κύριος Γιούρεκ, Γιούρεκ από τους Ευρωπαίους Συντατικούς Μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Α, θα είμαι σύντομα. Ε, θα αναφερθώ στο είπε ο κύριος Σαφχάουζερ. Ε, δεν ε, συμμερίζουμε τον τρόπο που ανέλησε τον πόλεμο στη Σορβία αλλά θα ήθελα επίσης να διαμαρτυρηθώ έναντι, σε σχέση με την ε, αντίδραση της πλειοψηφίας έναντι ε, νόμιμων μειοψηφιών. Αναφέρομαι στην ε, διακήρυξη ανεξαρτησίας του Κωσυφοποδίου που αμφισβητήθηκε από την Ισπανία. Αυτό υπήρξε το αντικείμενο μιας ανοιχτής συζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να παραμείνει αντικείμενο ανοιχτή συζήτηση στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Ο κύριος ε, Σταγιαννόφ, ε, πρωθυπουργός του Κόσοβο, διαμαρτυρήθηκε για τον πολλαπλασιασμό των χριστιανικών εκκλησιών στο Κωσυφοπαίδιο. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουμε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από, με την ε, μάχη έναντι των λεγόμενων εθνικισμών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ράντος από το Άλντε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ είμαι ευγνώμων προς τον συνάδελφο κύριο Βάγκελ, ο οποίος συμπεριέλαβε το θέμα αυτό στην ε, ημερήσια διάταξη. Επιτρέψατε μου καταρχήν να επισημάνω πόσο ανησυχητική είναι η κατάσταση σε, πολλές, σε σχέση με πολλές δηλώσεις που ακούστηκαν πρόσφατα. Ε, όπως ξέρετε, σήμερα στις Βρυξέλλες έχουμε ένα νέο γύρο συζητήσεων μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας. Η Σερβία ήρθε εδώ λέγοντας ότι το... να σταματήσει το τρένο ήταν μια πρόκληση και όχι αποστολή του τρένου. Και η Σερβία είπε ότι είναι πρόθυμη να πάει σε πόλεμο εναντίον του Κόσεβο όπως έκανε και στην ε, Κροατία. Ε, ένας ε, σημαντικός προσκεκλημένος στις συνεδριάσεις της σερβικής κυβέρνησης είχε καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου στο Βούκοβαρ. Μπορείτε λοιπόν να αντιληφθείτε πώς μια τέτοια είδηση αντιμετωπίζεται εκεί. Έχουμε επίσης εκπροσώπους του Κωσυφοπαδίου που πάνε στην Αλβανία για διαβουλεύσεις. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι δεν είμαστε σε θέση να επιλύσουμε τα θέματα τα οποία καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Φαίνεται ότι η πολιτική βούληση είναι ανεπαρκής και Ενδεχομένως ε, υπάρχει μια νέα διαίρεση των σφαιρών επιρροής στα Δυτικά Βαλκάνια, έτσι όπως ε, είχαμε στη Γιάλτα, μόνο που δεν έχουμε πλέον την σοφία του Winston Churchill. Τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να παραμείνουν μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να ενισχύσουμε την παρουσία μας εκεί. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κούγκαν, ειδικό ε, εμπειρογνώμων για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Οι πρόσφατε εξελίξει στι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων προκαλούν ε, πραγματικές σοβαρές ανησυχίες για μα. Δεν πρόκειται να παριθμίσω όλα τα θέματα αυτά. Ε, θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω αυτή την συζήτηση. Τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα. Βλέπω ότι οι διμερεί θέματα δεν ε, κλέπουν στην περιοχή αυτή. Χρειάζονται μια πολύ ευαίσθητη πολιτική προσέγγιση, όχι μόνο για τους πολιτικούς της περιοχής αυτής, αλλά και για μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, όπως βλέπουμε στις κοινοβουλευτικέ εκθέσεις, ε, δεν ξέρω πώς η ενταξιακή λογική ε, τελικά προβάλλεται εναντί άλλων ε, θεμάτων. Ε, πρόσφατα η ενταξιακή διαδικασία έχει επιβραδυνθεί. Κύματα εθνικισμού και πολιτικού σκεπτικισμού που διατρέχουν την Ευρώπη έχουν φτάσει στα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν, θέλ, θα ήθελα να τονίσω μόνο αρνητικά θέματα. Ωστόσο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα επόμενα βήματα και να προσπαθήσουμε να κατευνάσουμε τις καταστάσεις και να συνδράμε τις ε, φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν μετασχηματιστική δύναμη στην περιοχή αυτή. Αν δούμε για παράδειγμα τη Σερβία, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο. Εκεί οι μεταρρυθμίσεις προχωρούν. Έχουμε τη δυνατότητα να πειράσουμε τις εξελίξεις σε πολλές χώρες της περιοχής αυτής. Μέλη του σώματος ε, ανέλαβαν δραστηριότητα για να ξεπεραστούν οι πολιτικές κρίσεις στην περιοχή, ε, στηρίζοντας τις μεταρρυθμίσεις και ε, θα πρέπει να δεσμευτούμε περισσότερα και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποστείλει το μήνυμα ότι η διεύρυνση παραμένει στην ημερήσια διάταξη και θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Αλλιώς αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή αυτή θα σηματοδοτήσουν την αρχή ε, δυσμενών εξελίξεων. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κούκαν. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Σόφκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, η σταθερότητα της νοτιοανατολικής Ευρώπης για άλλη μια φορά αμφισβητείται. Υπάρχουν εντάσεις στη Βοσνία Ριζεχοβίνη, στην Σερβία, στο Κοσφοπέδιο και στη Μακεδονία, λέει ο Μιλήτρια τα θέματα για τη Ρεπόμπλικα Σέρψκα δεν είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και αυτά αντανακλώνται πάρα πολύ και από τη δική μου την προοπτική, από τα δημόσια μηνύματα που στέλνονται από τη Σερβία και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη προς μια ευρωπαϊκή χώρα, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κροατία. Υπάρχουν επιθέσεις κατά της Κροατίας από τη Σερβία, σε μεγάλο βαθμό σχετίζονται με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αλλά υπάρχουν και άλλα κίνητρα. Ο Υπουργό Εξωτερικών τη Κροατία το Δεκέμβριο ε, προειδοποίησε τι σερβικέ αρχέ ότι χρησιμοποιούν γλώσσα και εντάσει που ακούσαμε μόνο από το Μιλόσεβιτ στη δεκαετία του 90. Υπήρχε και επιστολή από τον κύριο Γιούνκερ προς τον κύριο Βούτσιτ για να ε, κατευνάσει λίγο τους τόνους και ε, ήταν αρκετά επιτυχής. Υπάρχουν μεν κάποιες εντάσεις, αλλά θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Κοινοβούλιο να επιδείξουν αλληλεγγύη προς την Κροατία όσον αφορά αυτές τις ε, ρητορικέ που ε, πυροδοτούν ε, τη βία όπως έκανε και ο πρόεδρος Γιούνκερ. Ένα μέλος της κυβέρνησης της Βοσνίας Ερζεγοβίνης επιτέθηκε στην Κροατία ε, για την επιστροφή ε, μαχητών του Ισλαμικού κράτους ε, στην Ευρώπη και κυρίως προς τη Βοσνία Ερζεγοβίνη που είναι μία από τη χώρα που έχει τη μεγαλύτερη εξαγωγή εντός εισαγωγικών μελών του Ισλαμικού κράτους. Αυτά τα οποία ακούσαμε είναι ρητορικέ της δεκαετίας του 90 και είναι και τμήμα του εγγενούς φασισμού της Κροατίας, όπως μας είπανε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ακούστηκαν στους πολέμους πριν από χρόνια. Προσπαθούμε όλοι να μειώσουμε λίγο τους τόνους, να κατεβάσουμε τους τόνους και καταλαβαίνουμε ότι κάποια κράτη-μέλη, αν αυτές οι εντάσεις ε, ε, κορυφωθούν αντί να μειωθούν, ε, τότε τα πράγματα μπορεί να είναι αρνητικά για κάποιες χώρες σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Η Κροατία έχει μια γεωγραφική θέση που σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα ασφαλείας τα οποία σχετίζονται με τα σύνορά της με τη Βοσνία, Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και επίσης και τις θαλάσσιες οδούς. Θα πρέπει λοιπόν ε, επειδή ακριβώς υπάρχει κίνδυνος αστάθεια στις χώρες αυτές, να προσέξουμε το ζήτημα. Η Κροατία ανησυχεί για αστάθεια λόγω μεταναστευτικών ροών και Ισλαμικού κράτους. Ό,τι και να γίνει στην περιοχή θα πρέπει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ουδέτερος μεσολαβητή στη διαδικασία και να μην επιλέγει πλευρέ. Δεν υπάρχουν νικητέ και ιτημένοι. Αυτό ήταν ο κανόνα όταν άρχισε να διαλύεται η πρώην Ιουγκοσλαβία και όλοι οι διεθνεί παράγοντες σεβάστηκαν αυτή την προσέγγιση. Έκτοτε βέβαια κάποιοι έχουν απομακρυνθεί από αυτή την πολιτική, όπω για παράδειγμα η Ρωσία, η Τουρκία και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ε, για να έχουμε και ένα κατάλληλο μείγμα λίγο ομάδων, η κυρία, ο κύριος Σάλτας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Βάγκελ για αυτή τη συζήτηση. Είναι μόνον ένα βήμα Απέχουμε μόνο ένα βήμα από την ε, ρητορική του μίσους έως την ένοπλη σύραξη. Αυτό το βιώσαμε ήδη πριν από μερικές δεκαετίες. Και θα πρέπει πραγματικά να αναγνωρίσουμε έγκαιρα αυτά τα μηνύματα, ούτω ώστε να μην συμβεί κάτι το οποίο θα έχει τραγικές συνέπειες. Ε, ρητορική μίσους, ε, ε, υποδάβληση ε, πολέμου. Όλα αυτά είναι εργαλεία του λαϊκισμού. Ο λαϊκισμός χρειάζεται βεβαίως και τους αντιπάλους του για να μπορέσει να αμφίσει. Ε, και όλα αυτά θα μπορούσαν να ρίξουν τις χώρες της της Βαλκανικής τεράστιες αναταραχές. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, αντιδράσουμε εγκαίρως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενισχύσει εδώ το ρόλο του, ιδιαίτερως όσον αφορά την υποστήριξη της, ε, του διαλόγου, ε, της ανεξιθρησκείας και της ανοχής γιατί ε, θα μπορούσαν τα περιστατικά αυτά να αυξήσουν τη δυσάρεστη αίσθηση ότι η κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια θα μπορούσε ενδεχομένω να κλιμακωθεί. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα χώρο διαλόγου και θα έπρεπε να υπάρξει δυνατότητα Αμοιβέ ανταλλαγής και προσπάθειες αναζήτησης λύσεων και με τους εκπροσώπους της Σερβίας και της ε, Μακεδονίας οι οποίοι δεν έχουν λύσει τα προβλήματά τους καθώς και με τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη αλλά και με εκπροσώπους της Ρεπούμπλικα Σέρψικα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να αποτελεί το χώρο ε, του διαλόγου και κατευναυσμού της κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τους Σλοβαίνους ομιλητές, ο κύριος Πίταρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα... Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και χαίρομαι που όλοι συμφωνούμε για τη βαρύτητα αυτής της συζήτησης. Πρόκειται για ένα στρατηγικό ζήτημα. Στο παρελθόν έγινε ένα συνέδριο στην Κροατία και τότε ε, θεματοποιήθηκε η ευρωπαϊκή προεπτική της ε, Κροατίας και μερικά χρόνια μετά ε, ελήφθη σχετική απόφαση. Ωστόσο τώρα το γεωπολιτικό πλαίσιο έχει αλλάξει. Δεν αναφερθήκαμε στην Τουρκία και άλλα συμφέροντα τα οποία συγκρούονται στην περιοχή αυτή. Πρόκειται για συμφέροντα τα οποία δεν ταυτίζονται πάντοτε με τα δικά μας ε, συμφέροντα. Ορισμένες πολιτικές ε, δυνάμεις ε, έχουν αποδειθεί σε ένα κυνήγι πολιτικών συμφερόντων και ακούγεται ο απόϊχος μιας ρητορικής μίσους ε, πάντοτε οι ίδιες ε, φράσεις, μια σύμμετρη εικόνα. Ε, σήμερα πηγαίνουμε με το σερβικό τρένο, αύριο κάπου αλλού. Νομίζω ότι ένα ψήφισμα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αρκεί σαν απόκριση σε όλα αυτά. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων προς τον κύριο Βάιγκελ που έθεσε το θέμα αυτό. Το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ειρήνης και να δώσουμε στις χώρες αυτές την προοπτική μιας ευρωπαϊκής ένταξης. Ε, μπορεί να θεωρήσουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι με τα όσα συμβαίνουν. Ε, θα πρέπει να αλλάξουμε κάτι, να αναθεωρήσουμε την πολιτική μας. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσει μια έντονη συζήτηση με την κυρία Μοργκερίνη, γιατί δεν είναι δυνατό να τερματιστεί η συζήτηση αυτή εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μποστινάρου τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση και θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος ε, και ε, συνεκτικός. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι αποτέλεσμα κάτι το οποίο γνωρίζουμε ευθύ εξ αρχή. Τα ε, συμπτώματα της κούρασης, της κόπωσης. Τα ιδρυτικά Βαλκάνια ήταν και θα είναι πάντα, εάν δεν δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρος αντιπαράθεσης ε, μεταξύ μεγάλων διεθνών παραγόντων. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία και τη γεωγραφία. Α, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι μπορούμε να κάνουμε στην πραγματικότητα πριν γίνουν οι χώρες της περιοχής ε, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να επενδύσουμε και σε υποδομές που βοηθούν τις χώρες να έχουν καλύτερη σύνδεση ε, είτε πρόκειται για οδικά δίκτυα, αυτοκινητοδρόμους, ε, σιδηροδρόμους και ε, αγωγούς φυσικού αερίου διαδρόμους φυσικού αερίου και επίσης θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την περιοχή να συμμετέχουν. Δεν αναφέρομαι στην περιφερειακή ιδιοκτησία, αλλά μια γενικότερη συνεισφορά και υποστήριξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της περιοχής, γνωρίζοντας ότι Ακόμα και πρόσφατα κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλαξαν την οτροπία της ε, για την περιοχή, κυρίως για διμερεί ζητήματα που συνήθως είναι είτε επίμαχα είτε ε, ζητήματα τα οποία οδηγούν σε ρήξη. Θα πρέπει λοιπόν αυτά να σταματήσουν. Και τέλος, φρονώ ότι είναι εξίσου σημαντικό να αναφέρουμε και την ανάγκη όλες οι χώρες οι οποίες ε, είναι σε διάλογο μαζί μας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να σταματήσουν να συμπεριφέρονται ε, με τρόπο ο οποίος αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Δεν μπορούμε να ε, κατονομάζουμε κάποιες χώρες απλώς και να λέμε ότι αυτοί είναι οι καλοί μαθητές και αυτοί είναι οι κακοί. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό και να ξεχάσουμε τέτοιες πολιτικές. Και τέλος, εάν συνεχίζουμε να αναβάλουμε αυτό το θεματολόγιο ε, και δεν παίρνουμε τόσο αποτελεσματικά βήματα, τότε κάποιοι άλλοι παράγοντες, η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία, θα είναι παρόντες στην περιοχή. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Η κυρία Πίτια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε προβληματίζομαι γιατί, και ανησυχώ γιατί η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ω προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων δεν είναι προδραστική. Ξέρουμε ότι τα Δυτικά Βαλκάνια αντιμετωπίζουν μία σειρά προκλήσεων και είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να εξακολουθήσουν να ακολουθούν τον δρόμο προς τη σταθερότητα και την ειρήνη. Δεν πρέπει λοιπόν να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά θα πρέπει με την ίδια προσέγγιση να αντιμετωπίζουμε όλε αυτέ τι χώρε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα μετρα και το σταθμό, θα ήθελα μόνο να αναφερθώ στη Μακεδονία. Η ομιλήτρια, όπω γνωρίζετε, ε, πληρούσε όλα τα κριτήρια για την ε, ένταξή τη και παρόλα αυτά την έχουμε αφήσει στον προθάλαμο εδώ και μια δεκαετία. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω όλα τα κρατημέλη μελη τη Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλου ε, να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με τη Μακεδονία. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι υπάρχει μια πιο ευνοϊκή προσέγγιση ως προς τη Σερβία, παρά το γεγονός ότι η Σερβία συνεχώς ε, ε, αποδεικνύει ότι δεν σέβεται τις ευρωπαϊκές αξίες. Και αυτό φαίνεται και από πρόσφατα παραδείγματα που οδήγησαν αυτές τις ε, εντάσεις στα Δυτικά Βαλκάνια. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και να διευκολύνει την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόβιν Μίκεν, επόμενος μιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πολωνικά για να είμαι όσο να το πιο ακριβής. Ελπίζω να με κατανοήσετε. Ε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς ε, φίλους ε, και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε τους σωστούς κανόνες και τις ευρωπαϊκές αξίες ή τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει όμως να, να, να ξεκαθαριστούν όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε τον κανόνα του εθνικισμού. Η κυρία Λούνατσεκ ε, επιτέθηκε στην αρχή του εθνικισμού. Όμως η κυρία Λούνατσεκ θυμάμαι ότι ήταν υπέρ της απόσχησης ε, της ε, Τσετσενίας. Γιατί να μην στηρίξετε λοιπόν και την απόσχηση της Κρυμαίας σε αυτή την περίπτωση. Η Σερβία δέχτηκε επίθεση γιατί ήταν κράτος πελάτης της Ρωσίας. Ε, όμως ε, το πρόσχημα για ε, το κοσμοπέδιο ήταν ο εθνικισμός. Έχουμε διαφορετικό εθνικισμό και και λαούς αν θέλετε εθνικότητες στη Σερβία. Για, εφόσον λοιπόν σέβεστε τον εθνικισμό, γιατί να μην δεχτείτε και το δικαίωμα της, ε, κάποιων περιοχών να προστεριστούν τη Σερβία ή αντίστοιχα με την Ρεπούμπλικα Σέρβσκα. Αποφασίστε τέλο πάντων, είστε υπέρ του εθνικισμού ή όχι. Τον αποδέχεστε. Ε, κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για την Καταλωνία. Αν σέβεστε τον εθνικισμό, θα πρέπει να σεβαστούμε και το δικαίωμα τη Καταλωνία να αποσχιστεί. Αναφέρατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση των χωρών. Να υπενθυμίσω ότι το 40% των χωρών σήμερα δεν αναγνωρίζουν το ανεξάρτητο κοσμοπέδιο. Ούτε η Ισπανία το αναγνωρίζει. Ισότιμη μεταχείριση λοιπόν απέναντι και σε αυτή την προσέγγιση, όπω και απέναντι στι χώρε που αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία του κοσμοπεδίου. Δεν είναι αλήθεια ότι όποιο ε, ε, καταφέρεται εναντίον τη ε, ανεξαρτησία του κοσμοπεδίου ε, δρά εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητώ λοιπόν ίση μεταχείριση. Ευχαριστώ κύριε Μικέ. Δεν θυμάμαι εγώ να μίλησα την Καταλωνία σήμερα το πρωί. ίσως ε, ήταν θέμα της διερμηνίας. Εγώ άκουσα αναφορά στην Καταλωνία. Τέλος πάντων, εφόσον ε, μιλάμε για την Καταλωνία, προφανώς και η Καταλωνία έχει το ίδιο δικαίωμα να αποσχιστεί από την Ισπανία. Εδώ δεχόμαστε και σεβόμαστε την εδαφική ακαιρεότητα όλων των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον τούτης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόκοβιτς είναι τελευταίος ομιλητής από το ΕΛΚ. Πού είναι. Ε, σας συγχαίρω για τον ε, διορισμό σας στη θέση αυτή ως Πρόεδρου. Υπάρχουν πολλοί μελητές από τη Σλοβενία. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε μετά την επίθεση στο Σεράγεβο. Σαν τη με την ε, Ευρώπη που 70 χρόνια μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο βρίσκεται στη θέση αυτή. Σήμερα η ιστορία της Ιουγκοσλαβίας εκτελήχθηκε διαφορετικά. Γνωρίζετε που οδήγησαν οι εθνικισμοί στη Ιουγκοσλαβία. Όπως ακούσαμε σήμερα, εκεί υπάρχουν πολλά αντικρουόμενα συμφέροντα ευρωπαϊκά συμφέροντα, συμφέροντα της ε, Ρωσίας, της Τουρκίας, άλλων μουσουλμανικών ε, χωρών. Και θα πρέπει και πάλι να πούμε ότι πολλοί ξένοι μαχητές προέρχονται από την ε, Βοσνία Ριζεγοβίνη Και αν δούμε τη σχέση μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας, βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν μεγάλες εντάσεις και στην ε, Μακεδονία υπάρχουν εντάσεις μεταξύ των ε, πολιτικών ομάδων και ε, με, τον και με, και με τα αλβανικά κόμματα, το αλβανικό κόμμα στην Μακεδονία. Εγώ υποστηρίζω την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δέσμευση των Ευρωπαίων να παρακολουθούν τις εξελίξεις στις χώρες αυτές. Γιατί εάν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, εάν εκλείψει η υποστήριξη εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα βαλκανικά κράτη δεν ε, θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Ε, εγώ υποστηρίζω αυτή τη διαδικασία και ελπίζω να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλη μετανάστευση από τις χώρες αυτές. Εάν ειρηνευθεί η περιοχή, τότε θα έχουν ένα μέλλον οι χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ και τώρα στο τέλος αυτής της συζήτησης θα ήθελα να δώσω το λόγο σε δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και από τη Γενική Διεύθυνση ΝΙΑΡ και θα ξεκινήσω με την κυρία Άσφωστ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και επιτρέψτε μου επί τη ευκαιρία να σας συγχαρώ και εσάς και τους αντιπροέδρους για την εκλογή σας εδώ σε αυτή την τόσο σημαντική επιτροπή και επίσης γιατί θέσατε τα Δυτικά Βαλκάνια ως πρώτο θέμα υπό την Προεδρία σας σήμερα. Βεβαίως η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι πολύ ανοιχτή σε συνεργασία με τα μέλη της Επιτροπής για όλα τα θέματα των Δυτικών Βαλκανίων, της Τουρκίας και όλα τα σχετικά ζητήματα που σας απασχολούν. Πάρα πολύ σημαντική συζήτηση, πάρα πολύ σημαντικά θέματα αναφέρθησαν και αυτό δείχνουν ε, τι όθηση δίνουμε και πάλι εκ νέου ως ε, συλλογική στρατηγική προσοχή προς την περιοχή. Η ύπατη εκπρόσωπος είπε ήδη από την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, συγγνώμη, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με τους Υπουργού Εξωτερικών ότι ε, πρέπει να εργαστούμε για τα Δυτικά Βαλκάνια για τους λόγους που ακούστηκαν και επίση αναφέρθηκε και ήδη ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων στην περιοχή εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ολοκλήρωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σημασία της Ευρώπης, τη σημασία της συμμετοχής στην οικογένεια. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η σημασία της ε, ανταλλαγής, ε, της άμεσης επαφής ε, και των πιο ε, τακτικών συζητήσεων, επισκέψεων και συνομιλιών είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό και είπα ότι εκπρόσωπος ζήτησε και πάλι να υπάρχει δέσμευση. Πρέπει να υπάρχουν οι διάφορες πλευρές και να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Υπήρξαν κάποιες επιτυχίες το 2016. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε και κάποιες ε, χώρες η ε, αίτηση συμμετοχή τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, το γεγονό ότι άνοιξαν κάποια νέα κεφάλαια με το Μαυροβούνιο και το Κωσυφοπαίδιο, τη δικαστική μεταρρύθμιση ε, ε, στις ε, εκλογές στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία και στο Μαυροβούνιο. όλα αυτά τα παρακολουθούμε και θα τα συνεχίσουμε να τα παρακολουθούμε το 2017 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα ενδιαφέρουν οι ευρωπαϊκές αξίες, να υπάρχει κατάλληλη προοπτική. Έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μα. έχουμε διάθεση και πλέον περισσότερο από ποτέ είναι προς το συμφόρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους ασφαλείας, εξωτερικής πολιτικής, σταθερότητας να εργαστούμε περισσότερο στην περιοχή. Και βεβαίως θα προωθήσουμε και όλα τα στοιχεία αυτά στις εργασίες μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Άσφολτς. Και τώρα η Κάθριν Ρέντ από τη Γενική Διευθυνσία. Εκεί είστε. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, και εγώ να σας συγχαρώ για τα νέα σας καθήκοντα και χαίρομαι για τη συνεργασία. Πολύ σύντομα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σαφώς και μας ανησυχούν οι πρόσφατες εξελίξεις και οι ρητορίες που ακούσαμε στην περιοχή. Έχουμε και κατά νου την προεκλογική περίοδο που πλησιάζει σε κάποιες από αυτές τις χώρες. Η περιφερειακή σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα παράδειγμα είναι η συζήτηση που έγινε προηγουμένως για τη μετανάστευση και το ρόλο που έχουν διαδραματίσει αρκετές χώρες στην περιοχή για να βοηθήσουν χρησιμοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ενισχύει και τη σημασία μιας σαφούς και απτής ε, προοπτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται και με τις χώρες αυτές και διμερώς και περιφερειακά ε, διαπραγματεύσεις σε διμερέ επίπεδο με το Μαυροβούνιο και το Κωσυφοπαίδιο συνεχίζονται. Ε, με τη Σερβία έχουμε συζητήσει τι πέντε βασικέ προτεραιότητε και ελπίζουμε να μπορέσουν να ξεκινήσουν ε, οι διαπραγματεύσει. και φυσικά μα ενδιαφέρει το θέμα τη μεταρρύθμισης του δικαστικού. Ε, η Βοσνία Ερζεγοβίνη έχει συζητήσεις, εξακολουθούμε να δούμε ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπως ανέφερε και η Αντζελίνα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη μετεκλογική περίοδο και στο Κωσυφοπέδιο η εισαγωγή του SAA είναι πολύ σημαντική βάση για τις μεταρρυθμίσεις με ε, κάποιο ευρωπαϊκό όραμα. Η διεθνή συνδρομή ε, σε οικονομικό επίπεδο συνεχίζεται και στα θέματα μετανάστευσης προς τη Σερβία και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας κυρίως. Και θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία και στα περιφερειακά στοιχεία τα οποία ε, προσπαθούμε να προωθήσουμε μέσω της διαδικασίας του Βερολίνου και την ε, συνεδρίαση των Βαλκανίων. Ε, στις 12 Ιουλίου θα έχουμε μια συνεδρίαση που ελπίζουμε ότι θα είναι πολύ σημαντικό ορότημα, ορόσημο και συνεχίζουμε για το θεματολόγιο για την νεολαία, το οποίο αναφέρθηκε η κυρία Λούνατσεκ προηγουμένως. Θέλουμε επίση να προωθήσουμε και θέματα δημόσια διπλωματία ε, με του συναδέλφου στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει προβολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι χώρε αυτέ για να υπενθυμίσουμε τι δεσμεύσει μα και να είναι βέβαιοι ότι θα τι υλοποιήσουμε. Ελπίζουμε ότι μπορέσουμε, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη δύσκολη κατάσταση με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε ψηφίσματα για τι πιο πρόσφατε εκθέσει σαν χώρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τη δέσμευσή σα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σε ευχαριστώ για... ευχαριστήσω για αυτή την πραγματικά πολύ εντατική συζήτηση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και του εκπροσώπου τη Επιτροπή. Θα ήθελα να κάνω τώρα τρει προτάσει. πρώτη. Ορισμένοι συνάδελφοι εξέφρασαν την επιθυμία να συνεχίσουμε τη συζήτηση για την κατάσταση στην περιοχή αυτή. Έτσι λοιπόν θα ρωτήσω, θα ζητήσω από τους συντονιστές. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε στην προσεχή μας συνεδρίαση να καλέσουμε τον Επίτροπο κύριο Χάνη την κυρία Μογκερίνη. Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ε, τη συζήτηση εδώ. Ε, θα έχουμε τις εκθέσεις για την εκθέσεις πρόοδο για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο και εγώ θα πάω στο Βελιγράδι και θα πω στους Σέρβους ε, εταίρους τα όσα άκουσα σήμερα από τους συναδέλφους των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Άρα θα έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα αυτά. Άρα λοιπόν θα ολοκληρώσουμε εδώ και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για τις ε, αξιόλογες εισφορές σας στο σημαντικό αυτό θέμα. Τώρα θα περάσουμε στο θέμα υπαριθμών 11. Νομίζω ότι οι Αιγύπτιοι συνάδελφοι και φίλοι έχουν ήδη μπει στην αίθουσα. Please take a seat next to me. Oh, hello, Ambassador. Good to see you. Good to see you. και μας φαίνεται So, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε τώρα στο σημείο για την Αίγυπτο. Θα ήθελα να χαιρετήσω θερμά εκ μέρους της Επιτροπής τον κύριο Αχμέτ Σαΐτ, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου. Κύριε Σαΐτ, καλώς ήρθατε στις Βρυξέλλες. Ε, επισκεφθεί επισκεφθήκατε τον περασμένο Απρίλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχατε συναντήσει με ορισμένα μέλη του σώματος. Ένα νέο κοινοβούλιο εξελέγει στην Αίγυπτο πριν από ένα χρόνο και εμείς βεβαίω θα ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη δική σας άποψη για τις πολιτικές ε, εξελίξεις ε, εντός της χώρας αλλά και περιφερειακά. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει το Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο, την κυβέρνηση και τα άλλα θεσμικά όργανα ε, προς την επίτευξη ε, πολιτικής σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί καλύτερη διακυβέρνηση, ιδιαίτερα όσον αφορά το χώρο της δικαιοσύνης και θα θέλαμε να ακούσουμε περισσότερα πράγματα για το καθεστώς ορισμένων νομικών εργαλείων, για παράδειγμα το νόμο για τις διαδηλώσεις και για τους νόμους για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Οι πρόσφατες αποφάσεις που ελήφθησαν από αιγυπτιακά δικαστήρια να παγώσουν ε, τα ε, δικαιώματα ορισμένων πολιτικών ακτιβιστών είναι ενισχυτικό στοιχείο. Πιστεύουμε ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι συστατικό στοιχείο της ημερούς μας σχέσης και θα θέλαμε να σας καλέσουμε να σεβαστείτε πλήρως τα, το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου. Επίσης θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις σας ε, εν σχέση με τον αυξανόμενο αριθμό δρομοκρατικών επιθέσεων στη Χερσόνησο του Σινά και την επίθεση κατά μια κοπτική εκκλησία στο Κάιρο. Θα θέλαμε να ακούσουμε επίση απόψει σας για την ε, εξέλιξη στην περιφέρεια και το ρόλο που διαδραματίζει η Αίγυπτο στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα όσον αφορά τη Συρία, την ε, Παλαιστινο-Ισραηλινή σύραξη και τη σχέση με τη Λιβύη. Ε, θα ήθελα να μας μιλήσετε για 10-15 λεπτά και στη συνέχεια θα έχουμε το χρόνο για μια συζήτηση. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να απευθυνθώ στα μέλη εδώ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και που μου δώσατε τη δυνατότητα να ρίξω κάποιο φω σε σχέση με το τι διαδραματίζεται στην Αίγυπτο. Επίση, θα ήθελα να δράξω μια άλλη ευκαιρία, την ευκαιρία αυτή για να συγχαρώ τον Ντέιβιν Μακάλιστερ για τον, την εκλογή του ως ε, καινούριο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εξωτερικών Υποθέσεων και πραγματικά χαίρομαι που θα συνεργαστώ μαζί του. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Έλμαρ Μπρόκ και όλες τις προσπάθειες και τη συμβολή του τα περασμένα χρόνια γιατί και η τελευταία του επίσκεψη πραγματικά εκτιμήθηκε πάρα πολύ στην ε, Αίγυπτο. Και καθώς ε, θα γνωρίσετε τελευταία έξι έτη η Αίγυπτος είχε αντιμετωπίσει μείζονες προκλήσεις. Ε, γιατί πριν από έξι χρόνια οι Αιγύπτιοι κατέβηκαν στους δρόμους ε, και είχαμε την, μια πραγματική επανάσταση προκειμένου να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, ε, οι ριζοσπαστικοί Ισλαμιστές ανέλαβαν την εξουσία. Παρ' όλα αυτά έχουμε ελπίδα, έχουμε ελπίδες Εν ώψη αυτής της κατάστασης, ε, τον Ιούλιο του 2014 οι Αιγύπτιοι και πάλι πήγαν, κατέβηκαν στους δρόμους και έλαβε χώρα μια δεύτερη επανάσταση η οποία ε, ήταν μια επανάσταση ε, για να προκειμένου να ανατραπεί μάλλον μια ιδεολογία και όχι μια, και όχι μια κυβέρνηση να, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ταυτότητα της ε, Αιγύπτου η οποία υπονομεύεται από τους Ισλαμιστές. Ήταν μια κραυγή εκ μέρους όλων των πολιτών της Αιγύπτου ότι δεν θέλουν να αποδεχθούν την ανάμειξη θρησκείας στην πολιτική και υπήρξε μια δραματική στιγμή την οποία θα διατηρήσουν ε, τα ιστορικά βιβλία γιατί οι Αιγύπτιοι χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν ε, αυτό το οποίο ήδη επιθυμούν. Ε, αυτή τη στιγμή οι τρομοκράτες έκαναν κατά επανάληψη βίες επιθέσεις στο Σινά και στο Κάιρο. Ο Γενικός Εισαγγελέας, ο ίδιος δολοφονήθηκε, ε, μέρα μεσημέρι. η στόχη των τρομοκρατών είναι να πληρωθεί ένα, ένας βαρύς φόρος αίματος ε, όσον αφορά την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο τουρισμός έχει μειωθεί δραματικά, το ίδιο και οι εμπορικές συναλλαγές. Επιτρέψτε μου όμως σήμερα να μιλήσω για το μέλλον και να σας πω το πώς πιστεύω ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Θεωρώ τη συνάντηση αυτή ως ιδιαίτερως ε, ενδιαφέρουσα, όχι μόνο λόγω των κοινών ε, στοιχείων που έχουμε και τις παρόμοιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, αλλά κυρίως λόγω του γεγονότος ότι τα τελευταία έτη τόσο η Αίγυπτος όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν να αντιμετωπίσουν στρεβλές εικόνες και παραποιημένες διατρεβλημένες αντιλήψεις. Ε, βεβαίως ε, και, είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια προοπτική στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αιγύπτου. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε υπογραμμίζοντα ότι δεν αρνούμε ανησυχίε στο από τη πλευρά ούτε από τη δική μα, αλλά θα προσπαθήσω να φωτίσω το πλαίσιο εντό του οποίου λειτουργούμε και όπου πραγματικά θα ήταν προ όφελον όλων μα να προσπαθήσουμε να βρούμε μια κοινή βάση. Είναι δύσκολο να ξαναφέρουμε στη μνήμη την πρόσφατη ιστορία όταν η περιφέρεια τη Μέση Ανατολή έζησε τόσο ταραχώδει ε, εξελίξει. Τα τελευταία χρόνια έφεραν ε, μαζί του μια πληθώρα προκλήσεων που φαίνεται δύσκολο να αντιμετωπιστούν ε, παρόλο που ξεκίνησαν μια θεμητή κραυγή των πολιτών, η Αραβική Άνοιξη, τα, οι περαιτέρω εξελίξεις δεν ε, αντανακλούν πάντοτε την αρχική πρόθεση. Και έξι χρόνια μετά την έκρηξη αυτών των διαδηλώσεων, η εικόνα είναι μάλλον ζωφερή. Η κατάσταση στη Συρία και στη Λιβύα ε, και παρά τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας δεν φαίνεται να πλησιάζουμε προς μια πύληση των συγκρούσεων που ε, ε, έγιναν εκεί. Στη Συρία και στη Λιβύη ε, τα προβλήματα θα πρέπει να κατανοηθούν σε δύο επίπεδα. Στο άμεσο επίπεδο, με την άμεση επίπεδο του πολέμου στις κοινωνίες αυτές και την διάδοση της κρίσης στην περιοχή αυτή επίσης την ανάγκη να ανοικοδομηθούν οι κοινωνίες αυτές και να μπορέσουν να ξεπεράσουν τη φρίκη του πολέμου. Επίσης είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η καταστροφή του πολέμου σε ορισμένε περιοχέ τη Μέση Ανατολή δεν θα πρέπει να μα κάνει να λησμονούμε το χρό... τη χρόνια σύγκρουση ε, στην Παλαιστίνη, ε, μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ. Ε, ορισμένοι προσπάθησαν να την υποβαθμίσουν σε σχέση με άλλε συγκρούσει, αλλά θα ήθελα πραγματικά να καλέσω όποιον σκέφτεται με όρους αυτούς να αναθεωρήσει την ε, αντίληψη αυτή σαν ως ιδιαίτερος επικίνδυνη. Γιατί η σύγκρουση Ισραήλ-Παλαστίνης θα παραμείνει ε, βασική ε, και είναι μια βασική αιτία προσιλητισμού Ισλαμιστών μεταξύ των νέων. Το να ισχυριστούμε ότι δεν υπάρχει θα ήταν βαρύτατο σφάλμα. Εμείς συνεχίσουμε να πιστεύουμε στην Αίγυπτο ότι η σύγκρουση αυτή είναι η μήτρα όλων των περαιτέρω συγκρίσεων και αν δεν επιληθεί ε, θα συνεχίσει να αναφλέγεται η Μέση Ανατολή. Όπως είπε ο Τζον Κέρι, αναφερόμενο στη σημασία της λύσης των δύο χωρών όσο και να μας εντυπωσιάζουν τα σχόλια του κυρίου Κέρι που είχε σαν μουσική στα αυτιά των Αράβων πολιτών, ε, πιστεύουμε ότι ήταν πολύ αργά ε, δύο μέρες πριν ε, λήξει η θητεία του Προέδρου Ομπάμα. Η Αίγυπτος βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη περιοχή. Προσπαθούμε ε, να προγραμματίσουμε το μέλλον, αλλά είναι πολύ δύσκολο, γιατί συνεχώς έχουμε απειλές για την εθνική μας ασφάλεια. Ε, με πάνω από χίλια χιλιόμετρα σύνορα με την ε, Λιβύη, με την απειλή του, της διεθνούς νομοκρατίας μέσω του ISIS και των μαχητών της, είναι πολύ εύκολο να διοχετεύσουμε ε, τους πόρους μας, ανθρώπινους, ε, πολιτικούς, οικονομικούς, προς την ε, ε, ανάπτυξη της ε, σταθερότητας, της οικονομικής ευρωστίας. Προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, γιατί παρότι έχουμε πολύ ισχυρές απειλές, ε, δεν μας έχει σταματήσει αυτό από το να οριστικοποιήσουμε ένα ε, σύγχρονο σύνταγμα στην εκλογή Προέδρου και ενός Κοινοβουλίου ε, που δεν είχαμε έξι χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο, μετά τη σύστασή του, το τελευταίο χρόνο δηλαδή, προσπάθησε να καλύψει το χαμένο χρόνο, ε, υιοθετώντα νομοθεσία που είχε αποφύγει το Κοινοβούλιο στο παρελθόν. Για παράδειγμα, ε, σε ό,τι αφορά την δημόσια διοίκηση, ε, που αλλάζει τον τρόπο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, με βάση δηλαδή την αξιοκρατία τους πλέον, ε, νέο φορολογικό, Ε, που είναι πλέον πιο δίκαιο, το, το νόμο που προβλέπει τη δυνατότητα των χριστιανών να γύρουν εκκλησίες που παλιά ήταν ένα όνειρο θερινής νυχτός ή μια χάρη αλλά τώρα θεωρείται θεμελιώδες δικαίωμα όπως και οι μουσουλμάνοι έχουν το δικαίωμα να χτίζουν τα τζαμιά τους. Και υπάρχει, προβλέπεται και ένας νόμος για την διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις ε, ε, άμεσες ξένες επενδύσεις ιδίω μετά τι πρόσφατε εξελίξεις ε, σε ό,τι αφορά την Αιγυπτιακή Λύρα που έδωσε ε, έδαφος ε, στην μαύρη αγορά και ενθαρρύνει άσχημε οικονομικέ εξελίξεις. Τέλος, ο νόμος για την παράτυπη μετανάστευση, ο οποίος ορίζει σαφώς για πρώτη φορά το έγκλημα της διακίνησης ανθρώπων ε, αποτρέπει αυτά τα φαινόμενα και τιμωρεί όσους ε, διακινούν ανθρώπους, ενώ αντιμετωπίζει τον μετανάστη ως θύμα και όχι εγκληματία. Κυρίες και κύριοι, σε μια διαφορετική χρονική στιγμή ε, θα μπορούσα να μιλήσω περισσότερο για τις απίστευτες επιπτώσεις τρομοκρατίας και του φόβου στη χώρα μας. Να μην ξέρει κανείς πότε και πού θα είναι η επόμενη μάχη μας. Όμως η Ευρώπη γνωρίζει και θα πρέπει να κατανοεί τι σημαίνει αυτό. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω ε, τι σημαίνει τρομοκρατία για μια χώρα ή για έναν λαό ή τις πιέσεις που δημιουργεί ε, για τα οικονομικά μιας χώρας όταν ε, είναι διατριτά τα σύνορα μιας χώρας. Θεωρούμε ότι αντιμετωπίζουμε αντίστοιχες, παρόμοιες και πολύ πραγματικές απειλές. Και αν θέλουμε να κατανοήσουμε ε, τις πιέσεις ε, τις οποίες δέχονται οι κυβερνήσεις εξαιτίας ε, της ε, τρομοκρατίας ή του μεταναστευτικού, κατανοείτε κι εσείς ε, τι πιέσεις δεχόμαστε εμείς ως τμήμα αυτής της περιοχής. Πρέπει να ασκήσουμε καθοδηγητικό ρόλο ε, στην ευρύτερη περιοχή και η Ευρώπη έχει δώσει πολύ σημαντικά δείγματα γραφή σε ό,τι αφορά την συμφιλίωση των λαών. Η ιστορία μα καλεί και μα υποχρεώνει να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε ε, τα πιο σημαντικά και τις πιο μακροπρόθεσμες ε, επιπτώσεις της κατάστασης που έχουμε στη Μέση Ανατολή. Από αυτή την άποψη η Αίγυπτος είναι διατεθειμένη και ικανή να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της λύσης του προβλήματος. Ε, θεωρώ ότι υπάρχει η καλή πρόθεση, ε, αλλά δεν θα πρέπει να ε, μείνει μόνη της ούτε η Ευρώπη ούτε η Αίγυπτος. Πρέπει να βρούμε τις αιτίε και τις διαδικασίες με τις οποίες έχουν κάποιοι καταφέρει να ακολουθήσουν μόνο αντιπαραγωγικές μεθόδους και μάταιες. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω ότι είναι σημαντικό για την ε, ευρωστία της εταιρική μας σχέσης να εργαστούμε από κοινού για τα κοινά μας συμφέροντα. Στόχος μου σήμερα είναι να θέσουμε το πλαίσιο για αυτή τη συνεργασία, γιατί όταν εξετάζω την περιοχή δεν βλέπω μια εταιρική σχέση που να είναι πιο ε, ισχυρή και αποτελεσματική από αυτή της, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος είναι μια ε, αρχαία χώρα και έδωσε όντως ε, τα αρχαιότερα πολιτιστικά μνημεία στον κόσμο. Όμως έχει και τις αδυναμίες της. Σήμερα η κοινωνία μας ε, προσπαθεί να βρει ε, θεραπείες και λύσεις. Έχουμε ε, πολλούς που έχουν παρισφρήσει στην κοινωνία μας. Έχουμε μια εισβολή του, των σκοταδιστικών δυνάμεων της περιοχής μας και όσοι επισκέφθηκαν την Αίγυπτο πριν από δεκαετίες μπορούν σήμερα κατευθείαν να διαπιστώσουν ότι έχουμε σημαντικά προβλήματα, αντιμετωπίζουμε και πολεμούμε τρομοκράτες γιατί είναι πιο εύκολο και πιο φτηνό, γιατί αυτό έχουμε δυνατότητα να κάνουμε. Αλλά αξιότιμοι συνάδελφοι, η πραγματική πάλι θα πρέπει να είναι ε, απέναντι στους ε, δημιουργούς των τρομοκρατών αυτούς που δημιουργούν ε, την ε, φτώχεια, που ε, βάζουν στα μυαλά του κόσμου την ιδέα του μίσους γιατί αξιοποιούν τη μοναδική ελπίδα αυτών των ανθρώπων, τον παράδεισο. Ναι, οι τρομοκράτε πιστεύουν ότι θα πάνε στον παράδεισο και δυστυχώ το να του μεταπίσει κανεί είναι μια μακρά και δύσκολη διαδικασία. Η μάχη λοιπόν κατά των δημιουργών της τρομοκρατίας είναι μια προσπάθεια που, στην οποία πρέπει να συμβάλλουμε όλοι γιατί η τρομοκρατία δεν ε, γνωρίζει σύνορα. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η πάλι ποτέ δεν θα πετύχει από μόνη της αυτή τη στιγμή γιατί αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα και όχι τις αιτίε. Η αιτία είναι η άγνοια και η φτώχεια. Για να την αντιμετωπίσουμε, να την αντιπαλέψουμε χρειαζόμαστε βοήθεια, συνεργασία, ε, κονδύλια και όχι δάνεια. Χρειαζόμαστε οι δήμονες και όχι οι πολιτικούς αναλυτές. Χρειαζόμαστε... Ε, πρέπει να δώσουμε ένα ε, πραγματικό μέλλον στην Αίγυπτο αντί να αναγκάζουμε τους ανθρώπους να πηγαίνουν στην Ευρώπη από την επελπισία τους. Προσπαθούμε να τους εκπαιδεύουμε τους, ε, τους πολίτες μας ε, στην Αίγυπτο και όχι να τους στέλνουμε ε, σε καριδότσουφλα στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Χρειάζεται όμως η Αίγυπτος βοήθεια από εσάς, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την τρομοκρατία από μόνη της. Όταν είμαστε ασφαλείς από την τρομοκρατία και όταν επιστρέψουν οι τουρίστες μας και οι επενδυτές μας, σίγουρα θα είμαστε σε θέση να επικεντρωθούμε σε άλλες μεγάλες αξίες που τώρα δεν έχουμε την πολιτεία να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να σας απευθύνω το λόγο. Σας ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαΐντ. 15 λεπτά ακριβώς μιλήσατε πριν ξεκινήσει και η συζήτηση, να καλωσορίσουμε τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Ντάμπη, ε, και φυσικά και τον πρέσβη, τον κύριο Χίγα Φαζήρο, ο οποίος είναι γνωστός ε, συνομιλητής μας. Και τώρα φτάνουμε στις ερωτήσεις και στα σχόλια. 11 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο, 12. Σας παρακαλώ το πολύ δύο λεπτά, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να μιλήσουν και φυσικά θα θέλαμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ξεκινούμε με τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας για την Αίγυπτο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην κυρία Ματίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για την εκλογή σας. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Ήθελα να ε, τον κύριο Σαΐτ και τον κύριο Νταρβής για την παρουσία τους εδώ και αθώς επίσης και τις, ε, την υπόλοιπη αντιπροσωπεία και τον πρέσβη. Είχαμε την ευκαιρία να πάμε στην Αίγυπτο τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου του 2016. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ε, αντιπροσωπεία, γιατί ήταν η επίσημη, η πρώτη επίσημη αντιπροσωπεία μετά από έξι χρόνια. Επομένως ήταν πολύ σημαντική η παρουσία μας εκεί. Θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και την επόμενη Τετάρτη στην συνεδρίαση της Επιτροπής ΑΦΕΤ εδώ. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ λοιπόν. Ήθελα απλώς να σας καλωσορίσω και ε, πιστεύω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου ε, και θα έχουμε φυσικά και τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε όλα αυτά ενδελεχώς ε, την Τετάρτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκαμπριέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Κύριε Πρόεδρε Σαΐντ, καταρχάς επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την πολύ εύστοχη παρέμβασή σας και να πω ότι πιστεύω στην κοινοβουλευτική διπλωματία και έχουμε και τακτικές επαφές μαζί σας, επομένως ε, νομίζω ότι καταφέρνουμε αυτή η ε, κοινοβουλευτική διπλωματία να είναι όλο και πιο ισχυρή. Η Αίγυπτος είναι τέρος ε, ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα όχι μόνο στη Μεσόγειο αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ στην Ευρώπη, σε όλη την περιοχή. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο ζητήματα. Καταρχάς το θέμα των προσφύγων και των μεταναστών που φτάνουν στην Αίγυπτο ε, η πλειοψηφία των προσφύγων και οικονομικών μεταναστών που είναι παράτυποι είναι από τις αφρικανικές χώρες. Η ερώτησή μου είναι τι σχέσεις έχετε με τις χώρες αυτές και κυρίως τι γίνεται προκειμένου να καταπολεπίσετε τη διακίνηση ε, μεταναστών. Επίσης, ε, ευτυχώς η κυβέρνησή σας ενέκρινε ένα νέο νόμο που ποινικοποιεί τη διακίνηση τον Οκτώβριο και ελπίζω να εφαρμοστεί. Το δεύτερο θέμα είναι σε περιφερειακό επίπεδο. Όπω είπα προηγουμένω, είναι ζωτική σημασία η Αίγυπτο για τη σταθερότητα στη Μεσόγειο. Πώ βλέπετε, το ρόλο τη Αιγύπτου στην Ένωση για τη Μεσόγειο, δεδομένου ότι θα γίνει και συζήτηση για την Προεδρία σύντομα και κυρίω ε, μία ερώτηση για τη Λιβύη και τη διαχείριση των συνόρων. Πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε οι μειονότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν αμφισβητούν σε καμία περίπτωση την ε, ε, ε, δαφική ακαιρεότητα της Λιβύης θα μπορέσουν να βοηθήσουν για τη σταθεροποίηση της περιοχής. Ευχαριστώ τη Μαρία Γαμπριέλ. Ο κύριος Φρόιντ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ πολύτως ε, με μία από τις ε, δηλώσεις στην παρέμβασή σας όταν αναφερθήκατε στην Ισραηλο-Παλαιστινιακή σύγκρουση ως τη μητέρα όλων των συγκρούσεων. Πράγματι, αν μπορούσαμε να επιλύσουμε αυτό το θέμα, ε, πολλά από τα υπόλοιπα προβλήματα της Μέσης Ανατολής δεν θα υπήρχαν και θα ήταν η Μέση Ανατολή πιο ειρηνική από ό,τι στο παρελθόν. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να τίνει ευήκονους στην έκκλησή σας και να δεσμευθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον προκειμένου να γίνει όχι μόνο ο μεγαλύτερος χορηγός στην περιοχή, αλλά και ο μεγαλύτερος παράγων στην περιοχή. Και κυρίως, και με αυτό έρχομαι και στο επόμενο σχόλιο μου, όσον αφορά τον νέο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρετε ότι αυτή είναι η τέταρτη ημέρα της προεδρίας του και κατά την τρίτη ημέρα ήδη συνομίλησε με τον πρόεδρό σας. Και αναρωτιέμαι, δεν ξέρω κατά πόσον γνωρίζετε καθόλου τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο κυρίων, αλλά ε, θα ήθελα να ξέρω τι προσδοκίες έχετε για, από τον νέο Αμερικανό πρόεδρο και όσον αφορά την κατάσταση στην Αίγυπτο, αλλά και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τζέφρι Βανόρτεν στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Κύριε Σαΐντ, ε, είστε πρόσδεκτος, αναγνωρίζουμε τη σημασία της Αιγύπτου ως ε, την πιο πολυπληθή αραβική χώρα και ε, σε πολύ κομβική γεωστρατηγική θέση, με ισχυρούς δεσμούς με πολλές από τις χώρες μας και πολλούς από εμά ε, η ασφάλεια, η ευημερία της Αιγύπτου μας απασχολεί ιδιαίτερα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τις δεσμεύσεις του Πρόεδρου Αλσίση ε, στον τομέα αυτό. Και θα ήθελα να αναφερθώ και ε, στα όσα ακούστηκαν από την τελευταία παρέμβαση. Το ζήτημα Ισραήλ-Παλαιστίνης βεβαίως είναι κομβική σημασίας, αλλά δεν πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για τις προϋποθέσεις οι οποίες υποθάλπουν την τρομοκρατία σε πολλές αραβικές χώρες. Αν θέλετε, αυτή είναι μια ξεχωριστή συζήτηση, την οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε σε άλλη στιγμή. Έχω κάποιες ερωτήσεις για σας. Καταρχάς, σε ποιο βαθμό ε, θεωρείτε ότι η τρομοκρατία εξαρτάται από εξωτερικές πηγές ε, ριζοσπαστικοποίησης, όπλων ε, και χρηματοδότησης. Ε, είναι κατ' ουσίαν εσωτερικό ζήτημα για την Αίγυπτο. Και δεύτερον, Ποια είναι η άποψή σας για την επιστροφή της Ρωσίας στην περιοχή με δεσμεύσεις τώρα και συμμετοχή στη Συρία και στη Λιβύη. Πιστεύετε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα προκειμένου να βοηθήσουν τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάγγελ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ομιλία σας, ήταν πολύ ουσιαστική. Δεν ήταν μόνο... Δεν είχε μόνο το χαρακτήρα μιας φιλοφρόνησης. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για, τα... για την πεποίθησή σας ότι η εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επιφέρει αμοιβαία ωφέλη και να ωφελήσει επίσης τη σταθερότητα και την ειρήνη. Θα ήθελα να σας απευθύνω ένα συγκεκριμένο ερώτημα εν σχέση με τις επαφές που εμείς ε, υποτίθεται ότι έχουμε με τη Γάζα. Ποια είναι η παρούσα κατάσταση ε, όσον αφορά τη ράφα, την διέλευση των συνόρων στη ράφα. Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα για ε, ανθρώπινες επαφές που υποτίθεται ότι έχουν διευκολυνθεί αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, παρακολουθούμε την Αίγυπτο σαν μια από τις δημοκρατικές χώρες στην περιοχή αυτή και μας ενδιαφέρει η εξέλιξη της δημοκρατίας σας. Θα ήθελα να σας απευθύνω μια έκκληση να καταλάβετε επίσης, να κατανοήσετε την αντιπολίτευση και τα, τις χρήσιμες ε, επαφές που μπορεί να έχει η κυβέρνηση με την κοινωνία των πολιτών. Βεβαίω συμμερίζομαι την άποψή σας και τα ε, αισθήματά σας ε, όσον αφορά την ομιλία του Τζον Κέρι. Ινσαλά. Θα μπορούσε να αποτελεί δηλαδή μια ευχή για όλους μας. Η επόμενη ομιλήτρια ε, κυρία Μπίλερ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, θυμάμαι τον περασμένο Μάρτιο που είχατε έρθει εδώ. Συστήσαμε επίση την κατάσταση των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων και το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα ήθελα να σας θέσω ορισμένες ερωτήσεις που είχαμε θέσει και τότε. Ε, συμφωνήσαμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις περιστατικά βασανισμών στην Αίγυπτο και το Κοινοβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο βελτίωση της νομοθεσίας ε, για τα βασανιστήρια και για τις εξαφανίσεις πολιτών γιατί η παρούσα νομοθεσία δεν ανταποκρίνεται στα διεθνή standards και έστω και αν ε, η Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είπε ότι χρήση βελτιώσεων όσον αφορά τα βασανιστήρια ε, και παρόλα αυτά όμως ε, υφίστανται και τα βασανιστήρια και οι εξαφανίσεις. και θα ήθελα να μας πείτε πώς προχωρήσετε στη μεταρρύθμιση αυτής της νομοθεσίας. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους υπήρξαν τόσα πολλά περιστατικά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, μεταξύ εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και μαχητών των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μία πάταξη ε, βίαιη του κινήματος των ακτιβιστών τι θα γίνει σε σχέση με τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις, θα αλλάξει σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ιδιαίτερα κατασταλτικά μέτρα που αντιμετωπίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απαγόρευση ταξιδίου, ε, ε ασφαλιστικά μέτρα, πάγωμα λογαριασμών κλπ. Ε, όλα αυτά, προσωρινές κρατήσει, όλα αυτά είναι ε, πολύ ανησυχητικά. Θα είχα περισσότερες ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αργότερα. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Σαφσάουζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ξεπεράσω το χρόνο μου. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, κύριε Σαΐντ για την ομιλία σας. Ε, έκανε τη διασκέψη και ο κ. Βάγκελ. Πραγματικά μιλήσατε με πειθό. Ήσασταν ε, ε, πιστικός και είναι σημαντικό γιατί έχετε μια νόμιμη εξουσία. Θα πρέπει να επιδείξετε και την ανάλογη ισχύ για να καταπολεμήσετε την, ε, τον Ισλαμισμό και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Και είναι αλήθεια ότι ορισμένες φορές υπάρχουν κάποια προβλήματα στην Αίγυπτο με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά εμείς οι Ευρωπαίοι ε, θα έπρεπε να θέσουμε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την παρέμβασή μας στη Συρία και στη Λιβύη και ας μην ξεχνάμε επίσης την παρέμβασή μας στο, ε, την επέμβασή μας στο Ιράκ. Και έχω ένα ερώτημα να σας θέσω δεν σκέφτεσαι ότι, δεν συμφωνείτε ότι υπάρχει μια θαυμάσια ευκαιρία με τη νέα Αμερικανική Προεδρία, τον πρόεδρο Τραμπ, να δημιουργηθεί η Συμμαχία για την Ασφάλεια και την Ανάπτυξη μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαίτερο τη όσον αφορά τη Βόρεια Αφρική που είναι πραγματικά μια ζώνη αστάθειας πολεμώντας κοινά τόσο την τρομοκρατία και ταυτόχρονα προωθώντας με την υποστήριξη της Αμερικανικής κυβέρνησης αυτό το πραγματικό σχέδιο Marshall το οποίο έχει ανάγκη η Αφρική γιατί όπως υπογραμμίσατε ο Ισλαμισμός τρέφεται από την φτώχεια και τον αναλφαβητισμό. Σας ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστούμε. Έξι ομιλητέ έχουμε ακόμα. Ο κύριος μόνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον κύριο Σαΐντ που ήρθε εδώ. Για μας, ε, τουλάχιστον για μένα, η Αίγυπτος είναι χώρα κλειδί στον αραβικό κόσμο και στην περιοχή. Όταν ε, αναφερθήκατε στην περιοχή που βιώνει τόσο δύσκολες ε, στιγμές ε, και στη διαδικασία της Συρίας ή της Λιβύης. Δεν ξέρω σε ποια από τις δύο αναφέρω γιατί από ό,τι ξέρω ο στρατηγός Χάφτερ ήταν στο Κάιρο πριν από λίγες ημέρες και αυτό μας ανησυχεί και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ε, ως Ισπανό εμένα που είναι χώρα της Μεσογείου. Ε, κάποιοι συνάδελφοι σας ρώτησαν για τις προσδοκίες της ε, Αιγύπτου για την Ένωση για τη Μεσόγειο. Εχθές δε συνεδρίασε στη Βαρκελόνη. Θα ήθελα να σας πω δύο νέα. Ε, νομίζω ότι είχαμε θετικά νέα από την Αίγυπτο τους τελευταίους ε, μήνες. Ε, την υπογραφή του συμφώνου με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιτέλους, πολύ σημαντικό για το λαό της Αιγύπτου, και μια αλλαγή στην ομοθεσία που επιβαρύνει τις ποινές για τους υπόπτους ε, και για όσου έχουν διαπράξει σεξουαλικά εγκλήματα, γιατί ξέρω ότι υπήρχε ατιμορρησία στα θέματα αυτά. Είναι καλή η είδηση αυτή λοιπόν και θα πρέπει να χαιρόμαστε όλοι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για την οικονομία ε, στην Αίγυπτο, που είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει κάποια βελτίωση για τον τουρισμό, μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα ώστε να προσελκύσετε και πάλι τουρίστες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την οικονομία της Αιγύπτου. Και επίση, ε, πώ βλέπετε το γεγονός ότι ο πρόεδρος Αλσίση εχθές μίλησε με τον εκλογέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει κάποια συμφωνία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά υπάρχουν και αυτές οι ιδέες της νέας ε, κυβέρνησης να αλλάξει πρεσβεία στο Τελαβίβ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, το αν η αλλαγή από το Τελαβίβ στα Ιεροσόλυμα θα ε, σας ανησυχούσε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παντσέρη στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Σαΐντ που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Ξέρω ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μια σειρά από αντικειμενικές δυσκολίες και σε επίπεδο κοινωνικής ισότητας και σε επίπεδο τρομοκρατίας και είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια σημαντική χώρα όπως η Αίγυπτος να έχει σταθερότητα διότι είναι πολύ σημαντικό για το σύνολο της περιοχής και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτή τη σταθερότητα. Ωστόσο, ε, στην απαραίτητη αναζήτηση της σταθερότητας ε, δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να θυσιάσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εδώ υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει ε, πορεία η χώρα σας. Η σημερινή σας παρουσία βεβαίως είναι σημαντική και λόγω μιας συγκεκριμένη συγκυρίας. Αύριο ε, έχουμε την επέτειο ε, του εις του Τζίλιο Ρετζένη στη χώρα σας και δυστυχώς ακόμα δεν έχει λάμψει αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιστάσεις, πολύ δισταγμοί από πλευράς ε, των αρχών της χώρας σας. Και εγώ θεωρώ ότι η αναζήτηση της αλήθειας είναι πάρα πολύ σημαντική και για την εξομάλυνση των σχέσεων με την Αίγυπτο και από εσά σήμερα περιμένω να πείτε κάτι από αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Grazie. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιούρεκ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα και για όλες τις σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε. Θα ήθελα να θέσω τα εξή σε τρία ερωτήματα. Πρώτον, πώς έχει κατάσταση στη Χερσόνησο του Σινά. βλέπουμε πώς ε, η Αίγυπτος προσπαθεί να ε, καταπολεμήσει την δημοκρατία. Ξέρουμε ότι οι στρατιώτες χάνουν τη ζωή τους, αλλά πείτε μας ε, λίγα λόγια παραπάνω για το τι συμβαίνει στην περιοχή αυτή. Ένα άλλο θέμα. Βεβαίως, όλοι ξέρουμε πόσο Σημαντική είναι η εξέβριση της ειρήνης μεταξύ Ισραηλινών και ε, Παλαιστινιακών αρχών. Όμως εδώ υπάρχει και το θέμα των αρχών της Χαμάς ε, στην Γάζα, στη λωρίδα της Γάζας. Είναι πρόβλημα νομίζω Χαμάς και για την Αίγυπτο. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τη δική σας εκτίμηση της κατάστασης σε ό,τι αφορά τα ανθρωπινά δικαιώματα στη λωρίδα της Γάζας. Υπάρχει κάποια πιθανότητα να αλλάξουν τα πράγματα εκεί, γιατί προς το παρόν εγώ δεν βλέπω κάποια προοπτική δημοκρατικής αλλαγής εκεί. Ίσως όμως ε, εσείς ε, να είστε πιο ενήμερος. Και το τρίτο θέμα που ήθελα να αναφέρω, η προοπτική της ειρήνης ε, στη Συρία. Πώς θα σταματήσει επιτέλους αυτός ο πόλεμος στη Συρία. Ευχαριστώ κύριος Πέτελε, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που βλέπω δύο νεοεκλεγέντες προέδρους ε, ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν ε, δράσεις. Καλή τύχη και στους ε, δύο. Κύριε Σαΐντ, ενθαρρυντικά τα όσα είπατε. Είπατε ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να μπλέκουμε τη θρησκεία με την πολιτική. Όντω μπορούμε να διαχωρίσουμε τη θρησκεία και την πολιτική θεσμικά, όμως δεν μπορούμε να ε, ξεχωρίσουμε τους πολίτες τους από τις ε, πεπιθήσεις και αξίες τους, που μπορεί να συνδέονται με τη θρησκεία είτε όχι. Θεωρείτε ότι ο διαχωρισμός ε, εκκλησίας κράτους θα ήταν χρήσιμο για την Αίγυπτο και πώς μπορείτε να εμβαθύνετε τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοβουλίων. Ευχαριστώ. κυρία Σλάιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε Σαΐτ, σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή. Ε, με πρόλαβε και ο συνάδελφος Παντσέρη. Αύριο είναι μια πολύ σημαντική επέτειος, η επέτειος ε, του χαμού του Τζίλιο Ρετζένη. Εσείς ζητάτε να προσπαθήσουμε τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου να τα βάλουμε σε μια σωστή προοπτική. Στη βάση όμως κάθε καλή σχέση υπάρχει ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη. Και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν μετά από ένα χρόνο να είμαστε ακόμα εδώ και να ζητάμε την αλήθεια. Εδώ υποδεχτήκαμε τους γονείς του Τζούλιου που είναι υπόδειγμα πολιτών γιατί έχουν μια διάκοπτη ε, ανάγκη για την αναζήτηση της αλήθειας. Υπάρχουν και πολλοί ακτιβιτές και πολίτες που ζητούν το ίδιο. Ζητάμε την αλήθεια για τον Τζούλιο. Γιατί πέθανε, ποιος το διέταξε, ποιος εκτέλεσε την εντολή και ποιος ε, ε, συγκάλυψε εννέα ημέρες βασανισμού και δολοφονίας ενός νέου ε, Ευρωπαίου ερευνητή. Χωρίς αλήθεια, χωρίς ε, ε, σεβασμό, χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρχουν φιλικές σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. τελευταίο ομιλητή ο κύριο Μπούχνερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Σαΐτ που ήρθατε εδώ και σας ευχαριστούμε πολύ και για την ε, συμβολή σας που είναι αξιόλογη. Τονίσατε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου ε, επιθυμείται να εντατικοποιηθούν και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται την Αίγυπτο και η Αίγυπτο χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο που αυτή τη στιγμή υπάρχουν εδώ κάποιε δυσκολίε. Θα γνωρίζετε ότι στην εμπορική μα συμφωνία, τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, πάντοτε υπάρχει μια ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ ξεκινούν τα προβλήματα. Για παράδειγμα, ότι οι χριστιανοί ε, έχουν προβλήματα και στην ε, κεντρική Αίγυπτο και στη Βόρεια Αίγυπτο. Ή για παράδειγμα οι δίκες αυτές όπου καταδικάστηκαν σε θάνατο 500 άτομα όπου ενώ ορισμένοι κατηγορούμενοι δεν είχαν καν ε, νομική συμπαράσταση τη δυνατότητα να μιλήσουν στη δίκη. Εσύ λέτε ότι δεν θα εκτελεστούν, αλλά θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τους έξι εκτελεσθέντες που εκτελέστηκαν για εγκλήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να είχαν διαπράξει γιατί ήδη την εποχή εκείνη ήταν στη φυλακή. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω επίσης τον βαρδισμό ε, χωριών στο Βόρειο Σινά. Ε, Πήγουσα, παράκληση να αντιστραφεί εδώ η κατάσταση, να εξασφαλιστούν καλύτερες προϋποθέσεις γιατί όπως είπατε οι δύο χώρες χρειάζονται η μία την άλλη και αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, δόκτωρα Σαΐτ, έχετε τώρα 14 λεπτά στη διάθεσή σας, γιατί πρέπει να κλείσουμε ακριβώς στις 12.30. Ε, αντί να απαντήσω με μονομένα σε ερωτήματα, θα απαντήσω στις θεματικές ενότητες, ε, λέει ο Πρόεδρος Σαΐτ. Βεβαίως έχετε ε, το ελεύθερο να απαντήσετε όπως θέλετε, αλλά σε 14 λεπτά. Παρακαλώ. Και πάλι σας ευχαριστώ. Με εντυπωσιάζει η γνώση και το ενδιαφέρον σας στα ζητήματα της Αιγύπτου. Βέβαια, το ξέρω, γιατί εκπροσωπώ και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεν μπορούσα να έχω εδώ τον επικεφαλής της ε, ομάδας ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολλά από τα ερωτήματά θα μπορούσε να τα απαντήσει καλύτερα εκείνο, αλλά δεν μπορούσα να εδώ σήμερα. Θα είναι πολύ δύσκολο για μένα να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα ξεχωριστά. Θα απαντήσω λοιπόν ε, στις θεματικές ενότητες. Ανθρώπινα δικαιώματα για τον, την περίπτωση του Ρετζίνη, την παράτυπη μετανάστευση. Ό,τι μπορώ να σας πω στα επόμενα 13 λεπτά που με απομένουν. Πρώτα απ' όλα, εκτιμώ ιδιαίτερω ε, το και τη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο. Είναι πολύ δύσκολο ε, να απαντούμε ε, ερωτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένα περιστατικά και γεγονότα. Όταν είπα στην ομιλία μου ότι θέλω να προβάλλω τις ε, σχέσεις μας, εννοούσα ότι είναι πολύ σημαντικό ε, να μεταφέρω ε, τις εντυπώσεις των Αιγυπτίων σε σχέση με, τα, με την προσέγγιση και αντιμετώπιση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο βέβαια, γιατί δεν θα σας πω για πριν από 50 χρόνια, αλλά πριν από 10 χρόνια κάποια πράγματα ήταν ένα όνειρο θερινή νυχτό. Ε, τα δικαιώματα των γυναικών για παράδειγμα, την ε, ίση πληρωμή ανδρών και γυναικών. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα σε αυτό. Ε, ισότιμα κληρονομικά δικαιώματα, σημαντική πρόοδο. Ελευθερία έκφραση. Ναι, βεβαίω και υπάρχουν αδυναμίε. Και το είπα ξεκάθαρα στην εισήγησή μου ότι δεν ήρθα εδώ για να σας πω ότι είμαστε τέλειοι. Κανείς δεν είναι τέλειος. Σίγουρα έχουμε και εμείς πράγματα που θα πρέπει να βελτιώσουμε να καταργήσουμε. Και εγώ δεν εκπροσωπώ εδώ τον ε, πρόεδρο ε, ε, της Αιγύπτου. Εγώ εκπροσωπώ το Κάιρο. Πάντα προσπαθώ να ασκήσω πιέσει στην κυβέρνηση, προσπαθώ να καταλήξω στην ε, αλήθεια και για μια χώρα που ήταν χωρί κυβέρνηση για 4-5 χρόνια και είχαμε μια χαοτική κατάσταση με 14 ψηφίσματα ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη Αιγύπτου τα τελευταία χρόνια, όταν δεν είχαμε ούτε πρόεδρο ούτε κυβέρνηση. Ε, ούτε κοινοβούλιο. Τι προσπαθώ να πω. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και βέβαια αυτό παίρνει χρόνο. Πολλοί μίλησαν για την ελευθερία έκφρασης. Μπορώ να σας πω ότι η Αίγυπτος είναι η μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή που έχει πλήρη ε, και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και στα μέσα δικτύωσης. Κανείς δεν το σκέφτεται αυτό αν ένας εκδότης Εφημερίδα δεν θέλει ας πούμε να δημοσιεύσει ένα ε, άρθρο, την επόμενη μέρα ε, υπάρχει παντού στο διαδίκτυο αυτό το άρθρο, γιατί έτσι λειτουργούν τα πράγματα και σε εμά. Για εσά αυτό μπορεί να ακούγεται φυσιολογικό, αλλά για πηγαίνετε στην Τουρκία, στο Λίβανο, ε, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εκεί πολλέ πολλές διαδικτυακές είναι κλειστέ από οποιαδήποτε συγκρατική ανάλυση θα δείτε ότι μια χώρα ε, σαν την Αίγυπτο με σχεδόν 100 εκατομμύρια κατοίκους, τη μεγαλύτερη χώρα στην Μέση Ανατολή, να έχει όλη αυτή την ελευθερία έκφρασης και ως προς το διαδίκτυο, αυτό δείχνει και την ελευθερία ε, της οποία χαίρει και η νεολαία. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ε, κακό σχήμανα τα οποία θα πρέπει να αλλάξουμε, βεβαίως. Όμως να λέμε και τα πράγματα όπως έχουν και να λαμβάνουμε υπόψη και την κατάσταση στη χώρα. Για παράδειγμα, για την κατάσταση στις φυλακές. Είχαμε τον πρόεδρο του ε, Ιρλανδικού Κοινοβουλίου. Πριν από δύο εβδομάδες ήταν ε, στην Αίγυπτο. Ήταν ένας νέος Ιρλανδός ε, που βρισκόταν στη φυλακή ε, και ήθελε εκείνο να πάει να τον δει. Και νομίζω ότι μετά κάνει μια πολύ σωστή ε, δήλωση. Είπε ότι είναι πολύ καλή κατάσταση. Ε, συνάντησε και τον πρόεδρο που είπε ότι θα βελτιωθεί περαιτέρω η κατάσταση. Επομένως, δεν χρειάζεται να ε, ε, επιμένετε τόσο πολύ. Εκτιμώ βεβαίω το ενδιαφέρον σα, αλλά πρέπει να ακούσουμε και τον λαό τη Αιγύπτου. Δεν είμαστε τόσο πλούσια χώρα όσο οι υπόλοιπε χώρε του κόλπου. Έχουμε οικονομικά προβλήματα, αλλά έχουμε μεγάλο πολιτισμό. Πρέπει να του ακούσετε λοιπόν και του Αιγυπτίου, του διανοητέ τη χώρα μου. Αν μιλήσετε, για παράδειγμα, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο, στη Συρία, τον πόλεμο διαδιπροσώπων, στον οποίο θα αναφερθώ σε λίγο, ε, για τα όσα συνέβησαν στο Ιράκ, που ξαφνικά τα ξεχάσαμε όλα και δεν ακούστηκε ποτέ μια συγγνώμη που χάσαν εκατομμύρια άνθρωποι τη ζωή τους χωρίς λόγο, ε, χωρίς να υπάρχουν ε, όπλα μαζικής καταστροφής. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε μπροστά και να δούμε πού θέλουμε να πάμε. Δεν υπερασπίζουμε ε, σε καμία περίπτωση τα όσα συμβαίνουν στην Αίγυπτο. Ίσως υπάρχουν και προβλήματα για τις ε, εξαφανίσεις, για παράδειγμα. Για το Στρασβούργο που πήγα πέρσι. Ε, το συζητήσαμε. Ακούσαμε έναν αριθμό 5.000 ανθρώπων. Εγώ είχα έναν αριθμό για 1.200. Πολλοί από αυτούς ε, προέκυπταν από την ε, άτυπη παράτυπη μετανάστευση. Γιατί αυτοί δεν καταχωρίζονται, ε, όταν φεύγουν μάλλον και μεταναστεύουν παράνομα, δεν ε, καταγράφονται πουθενά, δεν το λένε στους γονείς τους. Και εγώ οφείλω να μεταφέρω και είμαι υπόλογος στην περιοχή μου πάνω και κυρίω, περισσότερο από ότι στην διεθνή κοινότητα. Αλλά νομίζω ότι υπήρξε μια υπερβολή στα αριθμητικά στοιχεία. Δεν προσπαθώ να βρω δικαιολογίε, όμω πρέπει να λέμε και τα πράγματα όσου έχουν. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά. Αντιμετωπίζουμε απειλέ από τη Λιβύη με χίλια χιλιόμετρα σύνορα. Ξέρετε ε, όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ε, ISIS Υπήρξε και βομβαρδισμό με Β52, όπως ξέρετε. Έχουμε πρόβλημα με το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν. Ε, μετά όσο συμβαίνουν στα Δική Αραβία και στην Ιεμένη, με τη λωρίδα της Γάζας και τη Χαμάς, που αποτελεί προέκταση των αδελφών μουσουλμάνων και μετά κάποιος με ρώτησε τώρα τι σκοπεύετε να κάνετε για την ε, σύγκρουση με το Ισραήλ. Μα τι περιμένετε να κάνουμε εμεί μια χώρα που δέχεται όλε αυτέ τι πιέσει σε συνδυασμό με οικονομικά προβλήματα, με τον τουρισμό που με ρωτήσατε επίση, Είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε εδώ μια χώρα με, με τα δύο τρίτα των μνημείων ε, του κόσμου, με τις καλύτερες παραλίες, τα καλύτερα τοπία, με 11 εκατομμύρια ε, τουρίστες και είχαμε στόχο 20 με 25 εκατομμύρια. Ξέρετε όμως πόσους είχαμε πέρσι. 3,8 εκατομμύρια. Όταν είχαμε βάλει στόχο 25 εκατομμύρια. Φαντάζεστε λοιπόν ότι το 25% των Αιγυπτίων εξαρτάται από τον τουρισμό, όλη η οικονομία μας ουσιαστικά, και δεν έχουμε τουρισμό. Μας λένε, ναι, θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Αλλά περιπτώντως, Έχουμε πολλά να αντιμετωπίσουμε. Ίσως ε, υπάρχουν και ελλείψεις και αδυναμίες, αλλά κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας και στο Κοινοβούλιο για να ασκήσουμε πιέσεις ε, στην κυβέρνηση. Δύο πράγματα που θα ήθελα να φέρω για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ αρχικά. Είναι ιδιάζουσα η κατάσταση γιατί είχαμε πολύ κακές σχέσεις από το 2000 και μετά επί George Bush. Και δυστυχώς δεν είναι πολύ καλές οι σχέσεις. Τελευταία επίσκεψη Αιγυπτίου Προέδρου στις ΗΠΑ το 2004. Έχουμε 13 χρόνια λοιπόν να επισκεφθεί Αιγύπτιος Πρόεδρος στις ΗΠΑ. Για να είμαι ειλικρινής, είμαστε αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά τον Ντόναλτ Τραμπ και δεν βασίζεται αυτό σε σοβαρές ε, αναλύσεις. Απλώς βασίζεται στη σκέψη ότι δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Έχουμε πατώσει σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ. Και ήδη πριν ε, καν αναλάβει καθήκοντα, είχε αρχίσει να αντιπαλεύει τα κακό στη χώρα του. Ε, και βλέπετε ήδη και τι έγινε με όλε αυτέ τι τα λοιπά. Αλλά είναι περίεργα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στι ΗΠΑ. Αλλά όντω υπήρξε ε, και συνομιλία μεταξύ του ε, Αμερικανού Προέδρου και του Αιγύπτου Προέδρου. Δεν ξέρω τι λεπτομέρειε, αλλά προγραμματίζεται να υπάρξει επίσκεψη τον επόμενο μήνα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θα συζητήσουν πώ θα καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και ο κύριο Τραμπ ανέφερε στην ομιλία του πώ θα αντιμετωπίσουμε το ριζοσπαστικό και τρομοκρατικό Ισλάμ, αλλά δεν είπε πώς. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ερωτηματικά για το τι ακριβώ θα κάνει ο κύριο Τραμπ. Ταυτόχρονα έχουμε Αμερικανό πρέσβη στην Αίγυπτο με πολύ χαμηλό προφίλ, δεν έχει επαφή με κανέναν. Εγώ από τότε που είμαι πρόεδρο τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχω συναντηθεί σχεδόν με όλου του ε, πρέσβει ε, στην Αίγυπτο εκτό από τον Αμερικανό. Γιατί δεν ε, θέλει να φανεί. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα εξελιχθεί αυτό. Μετά, ζητήματα για τη Λιβύη, για τη Συρία. Και όλα αυτά εξαρτώνται από τις ΗΠΑ. Η Αμερική παλιά έκανε ό,τι ήθελε από το 1991 και μετά. Με τον πρώτο και δεύτερο πόλεμο του κόλπου, τώρα έχουμε ένα νέο ε, παίκτη στην αγορά που είναι η Ρωσία. Έχουμε εξαιρετικέ σχέσει με τη Ρωσία πριν από τον ε, βομβαρδισμό του ρωσικού αεροσκάφου. και από τότε έχουν ε, αλλάξει. Δεν ξέρω αν θα πάνε τα πράγματα καλύτερα ή όχι. Δεν ξέρω αν η σχέση μεταξύ Προέδρων ε, Πούτιν και Τραμπ ε, πώς θα εξελιχθούν. Πιστεύω όμως ότι τους επόμενους τρεις μήνες θα δούμε πολλά να αλλάζουν ε, στο διεθνές προσκήνιο. Και πάλι λοιπόν ε, τονίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για μια χώρα σαν την Αίγυπτο με πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα, προσπαθεί να αντιμετωπίσει ε, τη ρίζα της τρομοκρατίας, να αλλάξει ε, τον, την κουλτούρα αυτή, την αιτία δηλαδή και όχι τα συμπτώματα. τον θρησκευτικό διάλογο. Ίσως δεν παρουσιάζουμε πολύ καλά αυτό που κάνουμε. Όμως ε, πολλά καλά συμβαίνουν και πολλά αλλάζουν. Γι' αυτό και σας καλώ να έρθετε να μας επισκεφτείτε, να ακούσετε και να δείτε τι συμβαίνει. Σίγουρα όμως υπάρχουν ελλείψει, αδυναμίες. Το Κοινοβούλιο εργάζεται πολύ σκληρά για να βελτιώσει την κατάσταση, ασκεί πιέσει ε, στον Πρόεδρο. Το Κοινοβούλιο ανέλαβε ε, καθήκοντα από πέρσι είχαμε μια κυβέρνηση που δεν, έκανε, δεν ήταν υπόλογη σε ένα κοινοβούλιο. Ε, ξαφνικά τώρα αναστατώνεται ο πρόεδρος όταν το κοινοβούλιο τον, ε, το ρωτάει να ενημερώσει για το ένα για το άλλο θέμα. Ε, είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει τεράστιο πληθωρισμό αυτή τη στιγμή. Έχουν διπλασιαστεί οι τιμές σε πολλά αγαθά. Προσπαθούμε να εισαγάγουμε νέο επενδυτικό νόμο που θα ε, προσελκύσει ε, επενδυτές. Ασκούμε πιέσεις στον τραπεζικό τομέα για να αλλάξει ε, την μέθοδο, την προσέγγιση που ακολουθεί, να χορηγεί δηλαδή δάνεια μόνο στους μεγάλους κετρανούς. Θέλουμε να δίνει και στους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες στην Αίγυπτο. όσον αφορά την υπόθεση του Τζούλιο Ρετζένη, πραγματικά είναι ένα από τα θέματα τα οποία με θλίβουν ιδιαίτερα, ένα από τα μεγάλα σοκ. Να πω στους Ιταλούς φίλους εδώ στην αίθουσα που ρώτησαν για αυτή την υπόθεση, αν πάτε στην Αίγυπτο και επισκεφτείτε την Αίγυπτο ε, και ε, καλέστε ένα ταξί να σας πάει στο, στο ξενοδοχείο σας και σας ποιο είναι το όνομα του Ιταλού ανθρώπου με τον οποίο υπάρχει πρόβλημα, θα σας πει τον Τζούλιο Ρετζένιο. Ακόμα και ο ταξιτζής το ξέρει. Αν πάτε σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και συζητήσετε το θέμα, όλοι γνωρίζουν την υπόθεση πολύ καλά. Όλοι γνωρίζουν ε, το όνομα αυτού του ανθρώπου. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία είναι αδιαβόητη στην Αίγυπτο και είναι δραματική και δύσκολη για όλους τους Αιγυπτίους. Δεν σας το λέω αυτό για να κερδίσω τη συμπάθειά σας. Προσπαθώ απλώ να σας διαβιβάσω το μήνυμα ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Αιγυπτίους, πολύ περισσότερο και από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Προσπαθώ να σας διαβιβάσω το μήνυμα ότι ο Αιγυπτιακός λαός πριν ε, ακόμα και από το Κοινοβούλιο πιέζουν. Αν δείτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πόσα άρθρα γράφονται, πόσες εκκλήσεις υπάρχουν για να μαθευτεί αλήθεια. Εγώ ως ε, βουλευτής, ε, οι τελευταίες ειδήσει βέβαια που έχω είναι ότι οι ερευνητές ε, ε, συναντήθηκαν, νομίζω ο Γενικό Εισαγγελέα επισκέφθηκε τη Ρώμη και υπήρχε και αντίστοιχη επίσκεψη και έγινε κάποια δήλωση από την Ιταλική κυβέρνηση και από το Γενικό Εισαγγελέα τη Ιταλίας στη Ρώμη ότι δεν ε, ε, ε, όχι ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά είναι ικανοποιημένοι με την πρόοδο και πιστεύουν ότι θα καταλήξουν σε συμπέρασμα σύντομα. Δεν ξέρω περισσότερα να σας πω, αλλά ξέρω ότι είναι και η επέτειος του θανάτου του αύριο. Ζητούμε συγγνώμη για αυτό το οποίο συνέβη, λυπούμαστε πολύ και δεν θα σιωπήσει η Αίγυπτος μέχρι να αποκαλυφθεί αλήθεια. Ξέρω ότι δεν έχω άλλο χρόνο, συγγνώμη που σας καθυστέρησα, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σαΐτ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που απαντήσατε όλες αυτές τις ερωτήσεις και τα θετικά σας σχόλια. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο Δόκτωρ Σαΐτ δεν είναι απλώς ένας επιφανής Αιγύπτιος επιχειρηματίας στον τομέα της πληροφορικής είναι επίση και η ηγετική πολιτική φυσιογνωμία σε αυτή την σημαντική χώρα. Με εξέπληξε όμω που διάβασα και ότι είστε και ιδιαίτερα επιτυχημένο κολυμβητή. Ε, ήσασταν αθλητή ε, στα νιάτα σα, και η κολυμβητική σα καριέρα ε, κορυφώθηκε με τη συμμετοχή σα στου Ολυμπιακού του Λος Άντζελες το 1984. Πολύ εντυπωσιακή καριέρα σα, λοιπόν, εντυπωσιακή προσωπικότητα. Σα ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για την πολιτική σα σταδιοδρομία σε μια χώρα που είναι τόσο σημαντική και τόσο κρίσιμη κρίσιμη για τη σταθερότητα στην περιοχή. Αγαπητέ συνάδελφοι, για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τους προσκεκλημένου μας από την Αίγυπτο και θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση στις 3 η ώρα με τον ε, Μαλτέζο Υπουργό Εξωτερικό, τον κύριο Τζόρτζ Βέλλα. Σα ευχαριστώ πολύ.